Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Σας χαιρετίζω ολόθερμα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού όπου καλωσορίζουμε επειδή έχουμε και περισσότερο χώρο για να τους καλωσορίσουμε πολυάριθμους ε, προσκεκλημένους λόγω βεβαίως της παρουσίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος Σίλβα Καλδέρα, τον οποίον χαιρετίζω ιδιαίτερα θερμά με τους συναδέλφους του. Είναι πάντα ένα σημαντικό γεγονός όταν μας παρουσιάζεται σε εμά, την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Την παρουσιάζεται λοιπόν και στο Κοινοβούλιο. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ένωσης, είμαστε άμεσα εκλεγμένοι, οπότε παρουσιάζουμε στους πολίτες την έκθεσή σας. Ε, χαιρετίζω επίσης ε, τον Επίτροπο Σεμέτα και τους συνεργάτες του. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα τυπικά της έναρξης της συνεδρίασης. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις. Όχι. Ωραία. Εγκρίνεται. Υπενθυμίζω ότι η συνεδρίασή μας είναι δημόσια η οποία ε, μεταδίδεται απευθείας ε, μέσω live stream. Υπάρχουν βεβαίως και καμπίνες διερμηνίας για να διευκολύνεται η εργασία μας. Επίσης, υπάρχει μία μελέτη ο κοινοβουλευτικό έλεγχο της εφαρμογή του προπολογισμού λέγεται η έκθεση. Αφορά λοιπόν την εκτέλεση του προπολογισμού. Η μελέτη αυτή είναι διαθέσιμη. Να σα υπενθυμίσω ότι αναφέρονται σημαντικά θέματα που μας ενδιαφέρουν, διότι στα πλαίσια της διαδικασίας ετήσιας χορήγησης απαλλαγής έχουμε ανάγκη από αυτή την πληροφόρηση για να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση. Αυτές ήταν οι εισαγωγικέ παρατηρήσεις από την πλευρά μου. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερής διάταξης, έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και να σας δώσω το λόγο, ε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Τσόιρα, κύριε Γκάερ, Επίτροπε μέτα αξιότιμα μέλη κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να παρουσιάζω στην Επιτροπή σας σήμερα την ετήσια έκθεση του συνεδρίου για την εκτέλεση του προπολισμού της Ένωσης για το οικονομικό του 2011. Ποιε είναι οι κύριε ε, παρατηρήσεις, τα κύρια συμπεράσματα. Οι λογαριασμοί για το 2011 παρουσιάζουν με σωστό τρόπο τα αποτελέσματα της λειτουργίας της και τι χρηματικέ ροέ στο τέλος του χρόνου. Το εισόδημα και η αναλήψη υποχρεώσεων δεν είχαν ουσιώδη σφάλματα. Ωστόσο, οι πληρωμές είχαν ουσιώδη σφάλματα με εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος 3,9% για το σύνολο του προπολογισμού. Αυτό το επίπεδο σφάλματος είναι παρόμοιο σε αυτό του 2010. Τότε ήταν 3,7%. Η έκθεση αυτή λοιπόν και το μήνυμά της είναι συνεπές με το μήνυμα των προηγουμένων ετών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μας εκπλήσει. Φέτος όμως έχει περισσότερη σημασία από ποτέ άλλοτε διότι τα δημοσιονομικά της Ευρώπης δέχονται σοβαρές πιέσεις. Πρέπει λοιπόν να δαπανούμε με πιο αποτελεσματικό και στόχο προσιλωμένο τρόπο τους πόρους μας. Διαπιστώσαμε πολλές περιπτώσεις όπου τα κονδύλια της Ένωσης είτε δεν χτύπησαν το στόχο τους, είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε παραδείγματα, για παράδειγμα, επιδοτήσεις ε, για εκτάσεις που δηλώθηκαν ω μόνιμοι βοσκότοποι, ενώ στην πραγματικότητα τμήματά του ήταν πυκνό δάσο. Μαθήματα επιμόρφωση για υπαλλήλου ε, πληροφορική που δόθηκαν και για άλλου υπαλλήλου. Δόθηκαν χρήματα για ένα κτίριο που ελέγεται ότι ήταν για γεωρική χρήση, ενώ δεν ήταν. Δήλωση δαπανών προσωπικού υπερβολικέ και αναπτυξιακή βοήθεια που κατόπιν δεν σεβάστηκε τον κανόνα καταγωγής για την αγορά εξοπλισμού και διαδικασίε σύναψη δημοσίων συμβάσεων που δεν ήταν ε, ορθά εφαρμοσμένε, αν και ορθά σχεδιασμένε. Όπω υποδηλώνουν τα παραδείγματα αυτά, το συνέδριο βρήκε σφάλματα πληρωμέ σε πολλά διαφορετικά προγράμματα και καθεστώτα δαπανών. Διαπιστώσαμε επίση ότι συνολικά τα συστήματα ελέγχου που εξετάσαμε ήταν μόνο μερικώ αποτελεσματικά. Δηλαδή, τα συστήματα ελέγχου δεν αξιοποιούσαν πλήρω το δυναμικό του για να αποτρέψουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα. Το συνέδριο κατέληξε ότι μόνο σε δύο τομεί, οι ε, ομάδες πολιτικής δεν υπήρχαν ουσιώδη σφάλματα το 2011. Είναι οι τομεί εξωτερικέ σχέσει, εξωτερική βοήθεια και διεύρυνση και διοικητικέ και λοιπέ δαπάνε. Στου ε, υπόλοιπου πέντε τομεί πολιτική είχαμε ουσιώδη σφάλματα, ιδιαίτερα αυτού που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιφερειακή πολιτική. Εκτιμούμε ότι το ποσοστό για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου περιβάλλον αλία και υγεία ήταν το πιο υψηλό και ήταν 7,7% το ποσοστό σφάλματος δηλαδή. Ενώ το εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος για την ομάδα πολιτικής περιφερειακή πολιτική ενέργεια και μεταφορές ήταν επίσης υψηλό, παρέμεινε υψηλό, ήταν 6%. Ακριβώς εδώ, σε αυτούς τους τομείς, διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη δέσμευση ότι θα υπάρξει έλεγχος από τις ε, εθνικές αρχές. Πρέπει να ελέγχουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τους ε, νοσιακούς πόρους, διότι οι εθνικές αρχές είναι οι φορείς που κάνουν την πρώτη προσπάθεια για να προστατεύσουν είναι στην πρώτη γραμμή της, προσπάθεια προσπάθειας προστασίας των πολιτών της Ένωσης. Είχαμε πολλές περιπτώσεις ανεπάρκειας των ελέγχων, αποτυχίας των ελέγχων. Πάνω από 60% των ε, ε, ελεγχθησών πράξεων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε από πλευρά των ε, εθνικών αρχών, στα πλαίσια των εθνικών αρχών, αρκετή πληροφόρηση για να διορθώσουν σφάλματα πριν ζητήσουν αποζημίωση από την Επιτροπή. Και επίσης διαπιστώσαμε ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι δεν γίνονταν σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε ένα κτίριο που δηλώθηκε ως αγροτικής χρήσης. Είναι παράδειγμα αυτό σφάλματος που δεν διορθώθηκε παρά το ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον οργανισμό πληρωμών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν τα σφάλματα μέσω αποτελεσματικότερης εφαρμογής των υφισταμένων συστημάτων αλλά υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωσης των συστημάτων, καθώς και βελτίωσης των ε, σχετικών καθεστώτων δαπανών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Υπάρχει και ανάγκη, αλλά υπάρχει και δυνατότητα να ενεργήσουμε τώρα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να, θεσμίσουν, να θεσπίσουν καλύτερους κανόνες και κατόπιν να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, βελτιώσει την εποπτεία της και να αξιοποιήσει ήδη τα πορίσματα από τις διορθώσεις που κάνει. Αλλά πρέπει να λαμβάνει αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο δαπάνησης των πόρων, των πόρων της Ένωσης, καθώς και για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις που, στις οποίες προβαίνουν. Μέχρι στιγμής έχω μιλήσει για το 80% περίπου των πόρων της Ένωσης που διαχειρίζουν τα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχει και ένα υπόλοιπο 20% που τελεί υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής όπου περιλαμβάνεται ο ζωτικό τομέα τη έρευνα. Η Επιτροπή, στα πλαίσια τη διαχείριση αυτή, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη συμμόρφωση με του όρου επιχορηγήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το συνέδριο κατέληξε ότι στον τομέα έρευνα και άλλε εσωτερικέ πολιτικέ είχαμε ουσιώδη σφάλματα. Θεωρούμε ότι για το 2011 ήταν γύρω στο 3% πολλά από τα σφάλματα και ε, αποτυχία των ελέγχων που διαπιστώσαμε ήταν παράλληλα και για τους τομείς συνδιαχείρισης. Κύρια, τομή, ε, κύρια πηγή σφαλμάτων ήταν υπερβολική δήλωση από τους δικαιούχους για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα πλαίσια έρευνας. Βάσει των ισιών των κανόνων, οι δηλώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου που να εκδίδουν ανεξάρτητες ελεγκτικές ε, εταιρείες αλλά στο 80% των σφαλμάτων που διαπιστώσαμε, παρά το ότι είχαμε θετικό πιστοποιητικό ελέγχου, διαπιστώσαμε σφάλματα λοιπόν. Επίσης διαπιστώσαμε ουσιώδη σφάλματα στις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές του τομέα εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικής βοήθειας και διεύρυνσης, που σε μεγάλο βαθμό είναι υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής. Επίσης διαπιστώσαμε σφάλματα στις πληρωμές που γίνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Επίση, η Επιτροπή έχει το καθήκον και την εφαρμογή του προπολογισμού τη Ένωση και μέσω τη υποβολή εκθέσεων για δημοσιονομική διαχείριση. Αυτό συμπεριλαμβάνει εκθέσει για την κανονικότητα των ε, συναλλαγών και τι επιδόσει που επετεύχθησαν. Επισημαίνουμε ότι κατά τη γνώμη των Γενικών Διευθυντών τη Επιτροπή, το εκτιθέμενο σε κίνδυνο παρατυπία ποσό αυξήθηκε από 0,4 δι ευρώ το 2010 σε 2 δι το 2011 αυτή η εκτίμηση είναι στην ουσία βελτίωση, γιατί αντανακλά το ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι στον τομέα της ανάπτυξης υπαίθρου, της συνοχής και της έρευνας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σφάλματος. Ωστόσο, το συνέδριο θεωρεί ότι η εκτίμηση αυτή είναι ίσως υποτίμηση, διότι μένει ένα υπόλοιπο ποσοστό σφάλματος και αυτό αποτελεί βάση εκτίμησης. Αυτό δεν ήταν ακόμη το 2011 αξιόπιστος δείκτης του βαθμού στον οποίο ε, υπάρχουν ε, ουσιώδη φάλματα ακόμη και μετά την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών. Οι εκθέσεις για τις επιδόσεις της Επιτροπής ε, καλύπτονται από το κεφάλαιο της έκθεσής μας που έχει τίτλο «Αποτελεσματικότητα του προπολογισμού της Ένωσης». Οι δύο βασικοί τρόποι με του οποίου η Επιτροπή λογοδοτεί σχετικά με τι επιδόσει είναι με τη νέα έκθεση αξιολόγηση των οικονομικών τη Ένωση, που βασίζεται στα επιτεχανόμενα αποτελέσματα και με τι αιτήσει εκθέσει δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων. Όπω ανέφερε και στην γνώμη του νωρίτερα φέτο στο συνέδριο, θεωρούμε ότι η πρώτη έκθεση αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2012 είχε μικρή προστιθέμενη αξία και συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν πώ αυτή η αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει πιο χρήσιμη για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των ε, κοινοτικών πόρων. Η Επιτροπή πρέπει επίση να βελτιώσει την ποιότητα των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων. Εξετάζοντα τι αιτήσει εκθέσει τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία και Ανάπτυξη Πέθρου, Περιφερειακή Πολιτική, Ανάπτυξη και Συνεργασία, το συνέδριο διαπίστωσε ότι οι δείκτες επιδόσεων θα μπορούσαν να συνδεθούν στην την επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, καμία από τις τρεις αυτές γενικές διευθύνσεις δεν παρουσίασε στοιχεία για τα ζητήματα της οικονομίας και τη αποτελεσματικότητα. Το κεφάλαιο που ε, αποκαλείται αποτελεσματικότητα του προπλισμού τη Ένωση περιλαμβάνει και πίσω ορισμένα διδάγματα από τι ειδικέ εκθέσει του συνεδρίου του 2011 για να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα. Προτείνουμε η Επιτροπή να χρησιμοποιεί ποιοτικέ εκτιμήσει αναγκών για να εκτιμά τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο τη πολιτική, να ορίσει στόχου πολιτική που θα διευκολύνουν την απόδειξη και κατάδειξη τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί και η ποιότητα αλλά και η έγκαιρη υποβολή στοιχείων. Κύριε Πρόεδρε, βελτιώθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο εξέτασης η δημοσιονομική διαχείριση. Αλλά πρέπει να κάνουμε αρκετά ακόμη μέχρι να φτάσουμε στο απαιτούμενο ύψος σε όλους τους τομείς οικονομικής διαχείρισης. Πολλά τα προβλήματα που καθορίσαμε στο παρελθόν εξακολουθούν, αν και σε μικρότερο βαθμό. Τα προβλήματα αυτά όμως σήμερα έχουν μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ. το γεγονό ότι μειώθηκε το ποσοστό σφαλμάτων κατά το συνέδριο αποδεικνύει ότι η βελτίωση των κανόνων και η βελτίωση του τρόπου σχεδιασμού των προγραμμάτων δαπάνηση μπορεί να βοηθήσει. Και τώρα με τις νομοθετικές προτάσεις για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και τα κύρια αίτια. Για πολλά χρόνια το συνέδριο έχει επίσης καλέσει για απλούστερους τρόπους δαπάνησης, σαφέστερους στόχους, πιο μετρήσιμα αποτελέσματα και πιο αποτελεσματικές ρυθμίσεις ελέγχου. Η ετήσια εκθεσή μας για το 2011 έχει επίσης πολλές συγκεκριμένες συστάσεις, όπως και οι γνωμοδοτήσεις που έχουμε ε, διατυπώσει. Οι γνωμοδοτήσεις μας περιλαμβάνουν επίσης παρατηρήσεις για τις νέες προκλήσεις για την οικονομική διαχείριση και την υποχρέωση λογοδοσίας. Όσον αφορά τις προτάσεις σχετικά με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, που θα καλύψει τους τομείς δαπανών που ενέχουν το μεγαλύτερο ενδεχόμενο σφάλματος, το συνέδριο εφιστά την προσοχή μας στην ανάγκη ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής, να βελτιωθούν οι μηχανισμοί διόρθωσης και ανάκτησης και να εξασφαλιστούν κατάλληλα συστήματα ελέγχου των χρηματοπιστωτικών μέσων. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, η καιρή είναι δύσκολη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικότερους κανόνες για τον τρόπο ε, εκταμίευσης των κονδυλίων της Ένωσης και τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους κανόνες. Με αυτόν τον τρόπο ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα αξιοποιηθεί καλύτερα, πιο αποτελεσματικά για να παράσχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας. Αυτό είναι το μήνυμα της ετήσιας έκθεσής μας που είχα την τιμή να σας παρουσιάσω σήμερα στην ουσία είναι ένα μήνυμα βελτίωσης της υποχρέωσης λογοδοσίας για τους κοινοτικούς πόρους. Είναι ένας στόχος που πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να πασχίσουν να επιτύχουν ένα στόχος που είναι στο κέντρο της στρατηγικής του συνεδρίου για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε Καλτέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την σαφέστατη σας παρουσίαση των κυρίων συμπερασμάτων της εκεί σας έκθεσής σας για την εφαρμογή χρήση του προϋπολογισμού του δημοσιονομικού έτους 2011. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού συγχαίρει το συνέδριο για την ετήσια του έκθεση που περιέχει τόσες σημαντικές πληροφορίες όπως το ακριβές ύψος του λάθους, ποσοστό του λάθους. Φαίνεται από εκεί όμως ότι δεν υπήρξαν σημαντικά λάθη ως προς τον ισολογισμό έσοδα-έξοδα και ότι τα λάθη που διαπιστώθηκαν ήταν ανάλογα και παρόμοια με εκείνα του 10 αν και λίγο αυξημένα. βασική πια, βασικό στοιχείο πληροφόρησης για μας είναι τέτοιου είδους εκθέσεις και χαιρετίζω το γεγονός ότι ακόμη μια φορά κάνετε και σύγκριση με προηγούμενους προϋπολογισμού προηγουμένων ετών για να υπολογίσετε το συνολικό ποσοστό λάθους. Συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν επίσης σε μερικές περιπτώσεις παρά την, το συγκεντρωτικό τρόπο με τον οποίο κάνουν τον έλεγχο δεν είναι ελεύθερα λαθών για την καλύτερη δυνατή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Επίσης συμφωνούμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν απλούστερους και αποτελεσματικότερους κανόνες όπως το ζητάει συνεχώς το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα δε η Επιτροπή μας κατά τις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές και κανονισμούς. Πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς όπως πρέπει, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο στοιχείο που πρέπει να λάβει υπόψη το Κοινοβούλιο ως προς τον δημοσιονομικό έλεγχο για την χρήση των ενωσιακών χρημάτων. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο μας χορηγεί μια σταθερή βάση για την τακτοποίηση των μεθόδων δαπάνησης των χρημάτων και μας δίνει και πληροφορίες για τη μέτρηση πιθανών προόδων. Έπειτα στο κεφάλαιο 10 της ετήσιας έκθεσης για δεύτερη φορά μιλάει το συνέδριο για αποτελεσματικότητα. Ξέρω ότι αυτό είναι καινούργια έννοια και πιο δύσκολο να περιγραφεί. Στην απόφαση απαλλαγή για το 10, η Κομισιόν ήδη είχε ένα κεφάλαιο που αφορούσε την αποτελεσματικότητα ή αποδοτικότητα της εφαρμογής του προϋπολογισμού που είναι το ίδιο σημαντική με την κανονικότητα. Και ίσως θα έπρεπε αυτή τη νέα προσέγγιση της αποδοτικότητας ή performance να την γενικεύσουμε για να υπάρχει καλύτερη μέτρηση των αποτελεσμάτων, θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και του οποίου η σημασία αυξάνεται συνεχώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να τονίσω τη σημασία που έχει για τους πολίτες η αξιολόγηση της καλής χρήσης του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ακριβώς αυτόν τον στόχο έχει να ελέγχει τον τρόπο δαπάνησης των κονδυλίων στις τακτικές αξιολογήσεις που κάνει και στους δημοσιονομικούς ελέγχους του για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων ενωσιακών προγραμμάτων. Έτσι προετοιμάζουμε το έδαφος για τον εξυγχρονισμό, για μεγαλύτερη κανονικότητα και λιγότερα λάθη όπως ζητάει και το ελεγκτικό συνέδριο για να καταλήξουμε έτσι σε ένα πρότυπο πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο όπως απαιτούν οι, τωρινές, οι τωρινοί κανόνες για τη δημόσια διοίκηση. Εδώ η Κομισιόν έχει και αυτή την ευθύνη της για τα αποτελέσματα που επιδεύτηκαν στη χρήση η εφαρμογή του προϋπολογισμού. Όσο για τις εκθέσεις της, για την αποδοτικότητα, το καλύπτει και αυτό το συνέδριο στο κεφάλαιο Getting Results που κάνει και ορισμένα, βγάζει και ορισμένα μαθήματα από προηγούμενες εκθέσεις και κάνει μερικές συστάσεις. Οι ειδικέ ε, εκθέσεις είναι βασική πληροφόρηση που χορηγεί η Κομισιόν στο συνέδριο και θα ήθελα να του ζητήσω να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και ακολουθώντας αυτή τη γραμμή για μια τέτοια ανάλυση σε περισσότερο βάθος για το κατά πόσον αποτελεσματικά γίνεται η χρήση, η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Πέρα από τα προφανή ωφέλη που θα έχει κάτι τέτοιο για την καλύτερη δυνατή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, θα μπορούσαμε έτσι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαστε και κοντινότερα στον πολίτη, κοντύτερα στον πολίτη αν ξέρουμε ακριβέστερα πόσο αποτελεσματικά γίνεται η χρήση του προβολισμού, δηλαδή των χρημάτων των. Σας ευχαριστώ κύριε Καλτέρα και σας και τους συνεργάτες σας για την παρουσίαση της έκθεσής σας και πριν δώσω το λόγο στους συζητητές μας, στον εισηγητή μας, θα ήθελα να ακούσουμε τον Επίτροπο Σέμετα για να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν για τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ορίστε κύριε Επίτροπέ μου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, κύριε Πρόεδρε Καλδέρα, αξιόλογα μέλη τη Επιτροπή και του Ελεκτικού Συνεδρίου, η δημοσίευση της έκθεσης έκθεσης ε, του Συνεδρίου είναι ακρογωνίω λήθο τη διαδικασία χορήγηση απαλλαγή για τον προπολογισμό. Οι συζητήσει στην Επιτροπή σα θα βασιστούν κυρίω στα απορίσματα και στι παρατηρήσει του συνεδρίου και στι απαντήσει που θα δώσει η Επιτροπή. Ε, είμαι ευγνώμων που μπορέσαμε να συνεχίσουμε το καλό πνεύμα συνεργασία που για άλλη μια φορά αποδείχθηκε σημαντική σταθερά στην παράδοση των σχέσεων μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής. Με τον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό που υιοθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα έχουμε μια σωστή και καινοτόμα βάση για την εφαρμογή της ε, τομεακής νομοθεσίας για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Ε, είμαι ευγνώμων που οι νομοθετικές αρχές κατέληξαν σε συμφωνία για αυτό το φιλόδοξο και αναγκαίο νομοθέτημα. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω την εισαγωγή της ετήσιας ε, διαχειριστικής δήλωσης για όλους τους συνδιαχειριζόμενους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σώματα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων σε επίπεδο κρατών μελών θα έχουν δυνατότητα να χορηγήσουν ουσιώδεις εγγύσεις και να αποδεχθούν την ανάγκη λογοδοσίας. Αυτό το μέσο εφαρμόζει συγκεκριμένα τι νέε υποχρεώσει επιτοπίων και λογιστικών ελέγχων των κρατών μελών για την εφαρμογή του προπολογισμού και τι ε, απορρέωσε ευθύνε που εισήχθησαν με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Περαιτέρω σημαντική εργασία για την επόμενη οικονομική περίοδο συνεχίζεται. Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω την πρωταρχική σημασία των νέων πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών και την ε, μελλοντική τομιακή νομοθεσία για να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει κάνει φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές προτάσεις που προωθούν την απλούστευση και την καλύτερη χρήση πόρων. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πολιτική συνοχή, όπου οι προτάσει τη Επιτροπή κάνουν καθαρέ δημοσιονομικέ διορθώσει των κανόνα, σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, ανοιχνεύσει εγκαίρω τι παρατυπίε. Η Επιτροπή καλεί του συνομοθέτε να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Πρόεδρό του για την ε, θαυμάσια συνεργασία μεταξύ, των, ε, μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και ελεγχόμενου. Το 2011 αποδεικνύεται ότι για άλλη μια φορά ότι προσθέτει αξία η έκθεση για την εφαρμογή του προπολογισμού, την εκτέλεση του προπολογισμού. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Καλτέρα, εκεί που λέει ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ τα δημόσια χρήματα πρέπει να σέβονται σωστές δημοσιονομικές αρχές. Να αναφερθώ σε μερικά από τα μηνύματα κλειδιά της ετήσιας έκθεσης όπως την παρουσίασε ο πρόεδρος Καλτέρα. Για πέμπτη συνεχή φορά το Ελληνικό Συνέδριο έδωσε ανεπιφύλακτη θετική γνώμη για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι διαπιστώνω ότι το λογιστικό μας σύστημα δίνει σταθερή και αξιόπιστη βάση για προετοιμασία των λογαριασμών μας εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε την ποιότητα και του υψηλού την υψηλού επίπεδου διαδικασία του λογιστικού πλαισίου μας. Μερικά σημεία κλειδιά του, των ετησίων λογαριασμών του 2011. Το 2011 το διαμεσονικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1,5 δις ευρώ. Αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που αποδεικνύει το υψηλό ποσοστό εφαρμογής των πιστώσεων πληρωμών για το 2011. Αν εξετάσουμε τον ισολογισμό, διαπιστώνουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των δανείων που δόθηκαν και των υπολείπων δανεισμού. Είναι δηλαδή 27,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίω στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έδωσε δάνεια κατά το 2011 στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για αντισταθμιστικές, αντισταθμιστικές ε, συναλλαγές, δεν έχουν αντίκτυπο στο οικονομικό αποτέλεσμα ή στο καθαρό ενεργητικό. Το κεφάλαιο για την προχρηματοδότηση αποδεικνύει μια συνολική αύξηση 1,5 δις. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα ποσοστά στα ποσά που έχουν να κάνουν με την κρατική βοήθεια που συμπεριλήφθη σε αυτό το κεφάλαιο για πρώτη φορά. Το επίπεδο της προχρηματοδότησης που διαχειρίζεται η Επιτροπή στην ουσία έχει μειωθεί κατά 700 εκατομμύρια. Οι τακτικέ καθαρίσει αυτών των πληρωμών, όπως προβλέπει ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμό, θα συμβάλλει σημαντικά σε περαιτέρω μείωση των κινδύνων. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει προσεκτικά την κατάσταση στον τομέα αυτό. Πριν περάσω τώρα στα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης αυτής του συνεδρίου όσον αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καντέρα και το συνέδριο, διότι διασφάλισαν συγκεκριμένα την συγκρισιμότητα των ποσοστών σφαλμάτων μεταξύ 11 και 10. Παρουσιάζοντας ένα συγκριτικό πίνακα στο σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης, το Συμβούλιο επιτρέπει στους αναγνώστες να δουν ποιες είναι οι τάσεις των ποσοστών σφαλμάτων ανακεφάλαιο. Παρά την νέα δομή και τις αλλαγές στη μεθοδολογία που εισήχθησαν για πρώτη φορά σε αυτή την έκθεση. Η Επιτροπή καλωσορίζει αυτά τα μέτρα και θα πρότεινε να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος παρουσίασης για τις επόμενες εκθέσεις, ούτω ώστε να έχουμε μια σταθερή δομή και για το μέλλον. Το συνολικό ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές το 2011 είναι λιγότερο από 4% και παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2010, όπως τονίζει και το συνέδριο στην έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 96% του προπολογισμού του 2011 είναι χωρίς φάλματα, χωρίς ουσιώδη φάλματα. Αυτό είναι θαρρυντικό. Όχι μόνο επιβεβαιώνει την συνεχή βελτίωση που σημειώσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά Λαμβάνοντα υπόψη επίση ότι αυτό το σταθερό αποτελέσμα επετεύχθη παρά το ότι ε, ο κίνδυνο για τι συναλλαγέ αυξήθηκε το 2011. Το ενδεχόμενο κίνδυνο. Όχι μόνο αυξήθηκε ο όγκο των πληρωμών, αλλά έγιναν πολύ περισσότερε ενδιάμεσε και τελικέ πληρωμέ που υπόκεινται σε πιο περίπλοκου κανόνε και συνθήκε και άρα πιο πολύ σε ενδεχόμενο σφάλματο. Επιπλέον, το 2011 το συνέδριο για πρώτη φορά έκανε ποσοτικές εκτιμήσεις για τις περιπτώσεις μη ε, ε, πολυμερούς συμμόρφωσης για ε, δικαιούχους της κοινή γεωργικής πολιτικής που αντι, αντι, αντι, αφορά το 0,1% του συνολικού σφάλματος 3,9%. Χάρη όμως στους ε, ελέγχους που έκανε η Επιτροπή μπόρεσε να ανακτήσει 1,84 δις ποσών που καταβλήθηκαν ε, λανθασμένα το 2011. Συνολικά, το συνολικό ποσό χρηματοπιστωτικών διορθώσεων και ανακτήσεων είναι γύρω στο 1,4% των πληρωμών του 2011. Αν ε, θέσουμε αυτό το ποσοστό σε σχέση με το συνολικό σφάλμα 3,9% που υπολόγισε το συνέδριο, θα δείτε ότι το καθαρό αποτέλεσμα των ε, ανακριβιών είναι πολύ κοντά στο όριο σημαντικότητας του 2% που χρησιμοποίησε και ο εξωτερικός ελεγκτής μας. Μία άλλη σημαντική αποτίμηση του συνεδρίου που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι τα προγράμματα που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη για τα προγράμματα αυτά οι παραβιάσει των εθνικών κανόνων είναι ένα σημαντικό τμήμα των συνολικών ε, σφαλμάτων. Για παράδειγμα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η σε βάθος ανάλυση μα ε, καταδεικνύει ότι οι παραβάσει εθνικών κανόνων αποτελούν το 86% του συνολικού ποσοστού σφάλματο. Αυτό σημαίνει ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1,9 από το 2,2 ποσοστό σφάλματος προέρχεται από παραβάσεις των εθνικών κανόνων. Αυτοί είναι κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη-μέλη. Οι δικαιούχοι στα κράτη-μέλη αυτά και οι εθνικοί φορείς πρέπει να ελέγχουν και να σέβονται τους κανόνες αυτούς. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο περίπλοκοι οι κανόνες και γι' αυτό έχουμε τόσα σφάλματα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά από κοινού. Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα απλούστευσης πέρυσι στα πλαίσια των πολιετών προοπτικών και των 57 κλαδικών προτάσεων. Ωστόσο, ο στόχος απλούστευσης ήδη σήμερα είναι κινδύνο. Στον πρώτο πίνακα επιδόσεων για την απλούστευση που υιοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαπιστώνουμε ότι ναι, μεν ε, σημειώθηκε πρόεδρος, για ε, πρόοδο συγγνώμη, ε, με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Οι προτάσεις που γίνονται κατά την τωρινή διαπραγμάτευση για την κλαδική νομική βάση προκαλούν σοβαρέ ανησυχίε. Για παράδειγμα, οι προτάσει ε, συμπεριλαμβάνουν δυσκίνητη διαδικασία λήψη αποφάσεων, πολύ βαριέ διαδικασίε γενικά, αδικαιολόγητα, για παράδειγμα, επιτροπολογία ή οι εφαρμοστικέ πράξει που αντικαθίστανται από ε, εξουσιοδότηση πράξη. Στον ε, τομέα κλειδί τη έρευνα, η Επιτροπή πρότεινε απλουστευμένου κανόνε συμμετοχή με βάση το πρόγραμμα Ορίζον 2020. Ο χρυσό κανόνα, ένα πρόγραμμα, ένα ποσοστό χρηματοδότηση, θέλει να διευκολύνει τη χρηματοδότηση. Στα ίδια πλαίσια, μία ενιαία πάγια χρηματοδότηση, δηλαδή ενιαίο πάγιο ποσοστό χρηματοδότηση για τα έμεσα στοιχεία του κόστους προβλέπεται, αλλά αυτές οι αρχές αυτή τη στιγμή ε, τίθενται ένα αμφιβόλο από τους νομοθέτες. Πρέπει όμω να κάνουμε περαιτέρω απλουστεύσει για να μειώσουμε το κίνδυνο σφάλματο. Τα κράτη-μέλη πρέπει και αυτά να κάνουν τη δουλειά του, να αντιμετωπίσουν την υπερβολική πολυπλοκότητα των εθνικών ρόλων, που οδηγούν σε λάθη από πλευρά των δικαιούχων και δεν επιτρέπουν ε, αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Αυτό είναι ένα μήνυμα που ήδη έχω ε, αποστείλει προς τα κράτη-μέλη όταν συζητήσαμε τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στο ΕΚΟΦΗΝ. Είναι ένα θέμα αυτό που όλο και περισσότερο προσέχουν οι ανώτατοι ελεγκτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να τονίσουμε επανειλημμένα ώστε να γίνει αντιληπτό. Παρακαλώ να το αποστείλετε στους συναδέλφους σας στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ας συνεχίσω τώρα με τα συμπεράσματα του ελέγχου του συνεδρίου το 2011. Όλες οι υποχρεώσεις και τα έσοδα για όλο τον προπολογισμό δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Όπως και οι πληρωμές για την εξωτερική βοήθεια, την ανάπτυξη, τη διεύρυνση και τις διοικητικές δαπάνες. Η κατάσταση στην πολιτική συνοχή έχει βελτιωθεί ουσιοδό από το 2010. Έχουν μειωθεί ουσιαστικά τα σφάλματα, το ποσοστό σφαλμάτων. Ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που για πρώτη φορά απέκτησε το δικό του κεφάλαιο στην έκθεση του συνεδρίου, η κατάσταση είναι πολλά υποσχόμενη. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, το ποσοστό σφάλματο μειώθηκε κατά 40% και το μεγαλύτερο ποσοστό των ε, λαθών που παραμένουν των σφαλμάτων οφείλονται σε σφάλματα στι δημόσιε συμβάσει. Αυτή η θετική εξέλιξη καταδεικνύει άλλη μια φορά ότι τα συστήματα ελέγχου και διαχείριση λειτουργούν πολύ καλύτερα για την τωρινή περίοδο σε σχέση με τι προηγούμενε. Επίση, καταδεικνύουν ότι η Επιτροπή επαγρυπνεί και είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα ε, νομικά εργαλεία στη διάθεσή τη, ούτω ώστε να, να διασφαλίσει τη σωστή χρήση των ε, ε, κοινοτικών πόρων και να σταματάει τι πληρωμέ μέχρι να ληφθούν οι αναγκαίε ενέργειε. Όμω τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν τι προσπάθειέ του να επιταχυνθεί η μείωση των σφαλμάτων σε αυτό το τομέα πολιτική, ιδιαίτερα διαπιστώνοντα αν γίνονται οι σωστέ επαληθεύσει τη διαχείριση, ούτω ώστε να προλαμβάνονται σφάλματα. Η αύξηση των σφαλμάτων στη Γεωργία Κυρίως αφορά την ανάπτυξη της Τα περισσότερα από τα σφάλματα στον τομέα αυτό έχουν να κάνουν με την επιλεξιμότητα των ε, προγραμμάτων επενδύσεων, τη δήλωση μη επιλεξίμου φόρου προς τη θέμενη αξία ή τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Γενικός Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης, Άγκρι, ήδη είχε προβλέψει αυτή την κατάσταση σε έναν βαθμό και εισήγαγε μια επιφύλαξη για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ετήσια έκθεση πολιτικής δραστηριότητα του 2011. Η επιφύλαξη αυτή συνοδεύτηκε από ενέργειες για να ε, διορθωθούν οι παρατυπίες και να προληφθεί η περαιτέρω σημείωσή τους κατά την ε, τρέχουσα και επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Κάναμε μια προσπάθεια να εκτιμήσουμε τις βασικές αιτίες των σφαλμάτων σε, σωστή σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών και τους οργανισμούς πληρωμών, ούτω ώστε να βρούμε και τα διορθωτικά μέτρα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Η πληροφόρηση και η συνειδητοποίηση στα πλαίσια των κρατών μελών αυξήθηκαν και το πρόγραμμα ελέγχου προσαρμόστηκε ούτω ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στο ποσοστό σφαλμάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε αυτή την κατάσταση η συμμετοχή των κρατών μελών και των αρχών των κρατών μελών πρέπει να ενισχυθεί. Πρόκειται για συνδιαχείριση. Οι εθνικοί κανόνε μπορεί να τίθενται εν κινδύνο. Ιδιαίτερα η συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών αρχών στην κατά την παράσταση διαδικασία του συνεδρίου απέδειξε ότι βοηθάει ιδιαίτερα για να εντοπιστούν προβλήματα στο επίπεδο των συστημάτων κρατών μελών ή όταν τίθεται θέμα εφαρμογή των εθνικών κανόνων. Γι' αυτό, σε αυτού του σωστά αιτιολογημένου τομεί και περιπτώσει, οι λεγόμενες τριμερείς συναντήσεις μπορούν να θεωρηθούν καλή πρακτική για να διευκρινίζονται τα θέματα και να ενισχύεται η αλληλοκατανόηση. Στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών έχουμε επίσης αύξηση του ποσοστού σφαλμάτων. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο τομέας πολιτικής είναι σωστό παράδειγμα του κυκλικού αποτελέσματος των προγραμμάτων, διότι οι πιο περίπλοκες πληρωμές γίνονται κυρίως προς το τέλος της ε, περίοδου αναφοράς. Η Επιτροπή εξετάζει τις περιπτώσεις και τις παρατηρήσεις του συνεδρίου, ούτω ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα Horizon 2020 θα οδηγήσει σε περαιτέρω απλούστευση, άρα λιγότερα σφάλματα. Ωστόσο, υπενθυμίζω ότι σφάλμα δεν σημαίνει απάτη. Σφάλμα δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν κάποιοι πόροι, χάθηκαν ή σπαταλήθηκαν. Σημαίνει ότι κάποια προγράμματα επηρεάστηκαν τη στιγμή που γινόντουσαν οι έλεγχοι του συνεδρίου από αδυναμίες στην εφαρμογή τους, όπως η δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού των δαπανών. Χαίρομαι, κυρίες και κύριοι, που το συνέδριο για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή τα πάει καλά. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω ότι η Επιτροπή θα πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που αναφέρει το συνέδριο. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την ανάπτυξη της υπαίθρου. Κάποιες από τις παρατηρήσεις του δικαστηρίου συνδέονται σαφώς με την επόμενη γενιά προγραμμάτων. Έχουν στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και δομή των κανόνων και προγραμμάτων που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν κατά την ε, τρέχουσα ε, περίοδο χρηματοδότηση. Η Επιτροπή γι' αυτό είναι δεσμευμένη να βελτιώσει το σχεδιασμό και τους κανόνες των προγραμμάτων σε διάφορους τομείς πολιτικής, ούτως ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, οι κανόνες, να διευκολύνει την ομότυπη πρόσβαση σε κοινοτική χρηματοδότηση, να μειώσουμε τα σφάλματα, να δώσουμε περισσότερη υπευθυνότητα Στου ε, εμπλεκόμενου φορεί, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη και περισσότερη διαφάνεια στα διχειριστικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή θα μπορέσει έτσι να έχει περισσότερα εργαλεία στην ε, διάθεσή τη για να παίξει καλύτερα τον υποπτικό ρόλο τη σε αυτό το τομέα συνδιαχείριση, στο ένα τομέα όπου, ε, που καλύπτει περίπου το 80% του προπολογισμού, όπου συνεργαζόμαστε με κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή προτείνει ότι όλε οι παρατυπίε που ανοιχνεύονται από την Επιτροπή ή το Συνέδριο και αφορούν Λογαριασμού που υποβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη πρέπει να οδηγούν σε καθαρέ χρηματικέ διορθώσει. Η Επιτροπή επίση θέλει να δώσει περισσότερη έμφαση στην αποδοτικότητα των προγραμμάτων μα και την προσθέμενη αξία που πρέπει να χορηγούν στου πολίτε και επιχειρήσει της χώρας μα. Ο προπολογισμό μα ε, έχει στόχο τις επενδύσει για του ε, λαού τη Ευρώπη και των εταίρων μα. Γι' αυτό οι καθαροί στόχοι και οι ε, δείκτες ε, ε, αποδοτικότητας κλειδιά περιλαμβάνονται, θα περιλαμβάνονται σε όλες τις προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι θα μπορέσουμε να μετρήσουμε την απόδοση, να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες και να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές πορείας. Ελπίζουμε οι νομοθετικές οι αρχές, οι αρχές που αποφασίζουν τις νομοθεσίες να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία ούτω ώστε η σημαντική προπαρασκευαστική εργασία για, ένα, για μια σωστή εφαρμογή να αρχίσει να μπορέσει να ξεκινήσει. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για να διευκολύνει όσο γίνεται καλύτερα την επερχόμενη συζήτηση για τη χορήγηση απαλλαγή για το 2010. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την ομιλία σας και για τα όσα μας είπατε για την Επιτροπή όσο προς την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στον φετινό εισηγητή για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, τον συνάδελφο Κόλινγκ Σκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Καλντέρα, κύριε Επιτροπέ Σομέτα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο σήμερα μας υπέβαλε ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχει το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Την ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προπολογισμού για το 2011. Για 18η φορά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ποσοστό σφαλμάτων. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό καταδεικνύει την ε, ευθύνη της Επιτροπής που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προπολογισμού αλλά και του Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ούτω ώστε οι πόροι των Ευρωπαίων φορολογουμένων ανδρών και γυναικών να δαπανώνται καλύτερα για να επιτυχάνονται οι στόχοι της Ένωσης. Η Επιτροπή σε αυτήν την νομοθετική περίοδο έχει ακόμη μια ευκαιρία να καταλήξει σε θετική αποτίμηση. Θα έπρεπε να μειωθεί στο ίμιση το ποσοστό σφαλμάτων κατά τη γνώμη μου. Και ε, με πολλή αγωνία θα ήθελα να δω αν θα επιτύχει αυτό το στόχο της ε, Κομισιόν. Αν εξετάσουμε τώρα τα πορίσματα αναλυτικότερα του συνεδρίου, θα διαπιστώσουμε ότι η εικόνα έχει κάποιες σκιές αλλά και φως σε ένα σημαντικό τομέα της εκτέλεσης του προπολογισμού όπου δαπανώνται πολλά χρήματα τον τομέα της περιφερειακής πολιτικής έχει μειωθεί το ποστό σφαλμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν βελτιώσεις, ότι πιάνουν οι προτάσει μας, πιάνουν οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, τις οποίες υποστηρίξαμε. Αρχίζουν τουλάχιστον να έχουν αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν σημαντικοί τομείς όπου το ποστό σφαλμάτων έχει αυξηθεί. Η γεωρική πολιτική και κυρίως η ανάπτυξη πέθρου, δηλαδή ο δεύτερος ε, πυλώνας και ο τομέας της έρευνα βεβαίω. Θα επανέλθω σε αυτό. Συνάδελφοι, είμαι σαφώς πεπισμένος ότι Πολύ εθνικοί προπολογισμού είναι αντικείμενο χειρότερη διαχείριση από τον δικό μα. Αλλά αυτό δεν είναι δική μα ευθύνη αποτίμηση. Αυτό είναι ευθύνη των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Δική μα ευθύνη είναι να ελέγξουμε τον προπολογισμό της Ένωσης. Και αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι ναι μεν ε, ε επισήμως, τυπικά, την ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή υπάρχει διαχείριση είναι σημαντική και η ευθύνη των κρατών μελών. Μπορούμε λοιπόν στρεφόμενοι προς το κτίριο Λήψιους, όπου μας λένε πολλά αυτές τις μέρες για καλύτερη δαπάνηση, στρεφόμενοι λοιπόν προς το κτίριο του Συμβουλίου, να πούμε αυτό που είπε ο πρόεδρος Καλτέρα, που θα ήταν σκόπιμο να τη λέμε συνέχεια, οι εθνικές αρχές κατά την διαχείριση και έλεγχο των κοινωτικών μέσων πρέπει να τα πάνε καλύτερα. Διότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους πολίτες. Είμαστε η πρώτη γραμμή άμυνας για τη σωστή διαχείριση των πόρων των πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς αποτιμήσατε διαβάζοντας την έκθεση. Εμένα σε ένα βαθμό με συντάραξε όταν διάβασε πόσο χαλαρή είναι η έλεγχη στο επίπεδο των κρατών μελών στην περιφερειακή πολιτική 60% των σφαλμάτων είχαν αναγνωριστεί ήδη από τα κράτη-μέλη. Εδώ διαπιστώνουμε ότι αυτό το σύνθημα καλύτερη δαπάνηση δεν πρέπει να έχει στόχο τις περικοπές, αλλά τους καλύτερους ελέγχους. Και αν τα κράτη-μέλη θέλουν να γίνεται καλύτερη δαπάνηση, better spending, γιατί δεν ε, κάνουν τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουν για να υπάρχει καλύτερη δαπάνηση. Γιατί το Συμβούλιο δεν το συζητάει εσωτερικά. Πώ τα πάνε τα κράτη-μέλη, μεμονωμένα. Πώ σέβονται τι δικέ του υποχρεώσει. Να έχουν συστήματα διαχειριστικών ελέγχων που να είναι σε θέση να δουν πώ δαπανώνται, εάν δαπανώνται κανονικά οι κοινωνικέ ε, χρηματοδοτήσει. Το Συμβούλιο, το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η έλεγχη αυτή είναι μόνο εν, κατά μέρο, εν μέρη αποτελεσματική. 60% όπως είπα των σφαλμάτων στην περιφερειακή πολιτική αναγνωρίστηκαν από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να ε, ε, συμπεράνω ότι το θέμα δεν είναι να γίνουν περικοπές. Το θέμα είναι οι δαπάνες να γίνονται με κανονικό τρόπο. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα από όσα έχουν κάνει μέχρι στιγμής και ίσως θα μπορούσαμε να παίξουμε και εμείς κάποιο ρόλο όταν θα συζητήσουμε ε, τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές 2014-2020. Στην περιφερική πολιτική βλέπουμε να έχει μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, ως απόλυτο ποσό εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλέ. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα δεν είναι επαρκή για να πάμε κάτω από το επίπεδο ουσιαστικότητας 2% και ξέρουμε πόσο ουσιαστική είναι η περιφερειακή πολιτική. Πρέπει λοιπόν να γίνει μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Θα πρότεινα λοιπόν να είναι στις συζητήσεις για την απαλλαγή που έχουμε ενώπιόν μας ένα από τα βασικά σημεία, ένα από τα κέντρα βάρους τι μπορούμε να κάνουμε για να οξύνουμε ακόμη περισσότερο σε παρέμβαση στους ελέγχους του 2008 που έχουμε, στο κείμενο που έχουμε ήδη το 2008, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε τα συστήματα ελέγχου και διαχείριση στα κράτη-μέλη. Να εξετάσουμε πώς γίνονται οι οικονομικές διορθώσεις αν μπορούν να γίνουν καλύτερα και νωρίτερα. Να θέσουμε απαιτήσει για τα νέα όργανα και αυτή τη νέα ε, ε, δήλωση ελέγχου από τα κράτη-μέλη. Ήδη ο προηγούμενος συζητητής, ο Κρίστοφερ Φέλνερ, είχε τονίσει ότι οι καθαρές διορθώσεις σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν τα σφάλματα πρέπει να γίνονται να έχουν οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ουσιαστικό εργαλείο και ο Επίτροπος ε, Σέμετα ανέφερε το θέμα του gold plating. Γιατί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να θεωρείται υπεύθυνη για ε, τα σφάλματα που, κάνουν τα κράτη-μέλη για τη χορήγηση των ε, δημοσίων συμβάσεων, για παράδειγμα. Είναι ένα θέμα ίσως λιγάκι προκλητικό, αλλά το θέτω. Γιατί αυτό το θέμα των πλακών χρυσού, gold plating, πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης, πρέπει να δούμε ποια από τα μέτρα αυτά μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Σε μερικές εβδομάδες θα συζητήσουμε με τον Επίτροπο Τσόλος, που όπως κάθε χρόνο συμμετέχει στην διαδικασία χορήγηση απαλλαγής για το δικό του τομέα αρμοδιότητας, όπως σημειώσαμε τώρα, τώρα περισσότερα λάθη. Γι' αυτό του ζητήσαμε προτάσεις για το πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η τάση. Και η πολιτική έρευνας. Είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση εδώ γιατί εδώ δεν έχουμε συνδιαχείριση. Η Επιτροπή για τον τομέα αυτό είναι αρμόδια και χαίρομαι που η Επίτροπος για τον τομέα αυτό είναι η πρώτη που θα έρθει εδώ στις συζητήσεις για την απαλλαγή, γιατί και από αυτήν αναμένουμε προτάσεις πώς οι διαπιστώσεις του συνεδρίου αποτιμώνται από εκείνην, τι έχει να πει για αυτές τις ε, προτάσεις ε, του συνεδρίου και τι θα κάνει η κυρία Γκεώργεν Κλίν για να μειωθούν τα σφάλματα σε αυτό το τομέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις τελευταίες δύο εκθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής, τουλάχιστον στις εσωτερικές συζητήσεις ε, αρχίσαμε να θέτουμε προτεραιότητες ενώπιον της Επιτροπής και απαιτούμε να εφαρμόζονται αυτές οι προτεραιότητες ούτως ώστε να μειωθούν τα, προγράμματα, τα ποσοστά σφάλματος. Οι δύο προηγούμενοι εισηγητέ, Χαζημαρκάκης και Φιέλνερ, ήδη ανέλαβαν αυτή την προσπάθεια, συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, να δείξουμε δηλαδή πρώτα απ' όλα σε τι βαθμό η Επιτροπή σεβάστηκε και εφήρμοσε τις προτεραιότητες των δύο προηγουμένων εισηγητών, τι έγιναν με τις εκθέσεις ε, συνέχισης, follow-up, και θα πρέπει και από την σημερινή έκθεση να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Έχω κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ποιες νέες προτεραιότητες θα πρέπει να θέσουμε, με βάση ακριβώς και τις επιπτώσεις από τις συζητήσεις ε, τις προπαρασκευαστικές για τη νέα δημοσιονομική περίοδο 14-20, αλλά και από τις προηγούμενες. Εδώ έχουμε μία ακόμη ευκαιρία για να έχουμε ουσιώδη μείωση των σφαλμάτων και να ανακτήσουμε τα ποσά των φορολογουμένων που δαπανήθηκαν λαθασμένα. Αυτή είναι η ουσία της εργασίας μας. Εδώ θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Γκάια. Ο συνάδελφο Γκάια εγγράφεται στην συνέχεια των προηγουμένων εισηγητών και της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου. Ανέφερε συγκεκριμένα θέματα η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από σημεία που πρέπει να συζητήσουμε και ήδη έχω μια σειρά συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, από πλευρά ΕΛΚ, ο συνάδελφος Μπίμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ε, χωρίς προβλήματα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκάια. Θα επιχειρήσω να αποφύγω επαναλήψεις. Όντως, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι διαφανής. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό τον κύριο Καλδέρα, τον πρόεδρο Καλδέρα. Είναι σαφής, εύκολα διαβάζεται, εύκολα την καταλαβαίνουμε, κατανέμεται σαφώς σε περιόδους. Εύκολα λοιπόν μπορούμε να διαμορφώσουμε εικόνα για τα θέματα που διακυβεύονται. Αυτό που μας ανησυχεί είναι το γεγονός ότι το 2009 ήταν ένα ναδύρ. Από τότε έχει βελτιωθεί η κατάσταση. 2010-2011. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει υψηλότερο ποσοστό σφάλματος. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς το το συνέδριο αυτό. Εδώ γίνονται κάποιες υποθέσεις. Γίνονται αναφορές βέβαια σε τομείς όπου έχουμε κυρίως σφάλματα. Ο Σάλφος Γκάερ αναφέρθηκε κυρίως στην πολιτική έρευνα Αυτό που με εξέπληξε εμένα, για μας μάλλον ήταν ε, αρκετά προσδόκητο, ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου είχε ποσοστό σφάλματος 7,7%. Πώς είναι δυνατόν σε αυτό το τομέα, όπου τουλάχιστον εγώ ξέρω τις διαδικασίες, είναι ιδιαίτερα διαφανής πώς είναι δυνατόν σε αυτό το τομέα να έχει ανέλθει, αυξηθεί τόσο πολύ το ποσοστό σφάλματος εδώ, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του συνεδρίου. Ακούσαμε ότι η ευθύνη είναι κυρίως ευθύνη των κρατών μελών. Ένα μεγάλο τμήμα της ευθύνης για τα σφάλματα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ε, νέα διαπραγμάτευση. Είμαστε σε αποφασιστική φάση νέων διαπραγματεύσεων για τα διευθυντικά ταμεία τι πορίσματα εξάγει λοιπόν από αυτήν την ευθύνη των κρατών μελών το συνέδριο για αυτέ τώρα τι επικείμενε διαπραγματεύσει για τα τα ταμεία και τα συστήματα ελέγχου. Τι αναμένεται ω βελτίωση. Κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τομεί, όπως οι δημόσιε συμβάσει, όπου βλέπω ότι γίνεται πολύ ισχυρή κριτική. Μιλάμε για την ε, αιρεσιμότητα. με βάση το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον, δηλαδή να περάσουμε περισσότερο σε εφαρμογή ενωσιακών και όχι εθνικών κανόνων για τη χορήγηση τέτοιων συμβάσεων. Τα κράτη-μέλη έχουν τις δικές τους ελεγκτικές αρχές στις οποίες αναθέτει τον έλεγχο. Και η Κομισιόν κάνει και το συνέδριο τον τελικό έλεγχο. Σε μια διαθροτική πολιτική η Επιτροπή όμως πρέπει να συμμετέχει πολύ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου και επιστοποίηση. Και ένα τελευταίο σημείο. Που εμένα με ανησύχησε ιδιαίτερα. Βλέπω κύριε Καλτέρα γράφεται εδώ ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας Περιφερικής Πολιτικής οι Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας Περιφερικής Πολιτικής και Συνεργασίας δεν ανέφεραν τις αρχές της ε, σωστής χρήσης πόρων. Αλλά 80% του προπολογισμού θα πανάται από αυτές τις ε, γενικές διευθύνσεις. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς. Βεβαίω αυτό το θέμα συνδέεται με τη στρατηγική 2020, με αυτού του δείκτε αποτελεσματικότητα στι διαστατικέ πολιτικέ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα βοηθήσει να υπάρχει σαφέστερη κατανόηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Αλλά αν δούμε αυτούς τους δείκτες, για παράδειγμα, τι ποσοστό παιδιών είναι σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, τι ποσοστό μαθητών εγκαταλείπει το σχολείο, Πού μας οδηγούν αυτοί οι δείκτες. Καλή προσπάθεια να δούμε ε, περισσότερο τι αποτέλεσμα έχουν οι πολιτικές μας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Γιατί μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Τέλος. Είπαμε ότι θα ακούσουμε τους επιτρόπους για να μας δώσουν τι απαντήσει που περιμένουμε για τους τομείς πολιτικής ε, για τους οποίους είναι αρμόδιοι. Το βασικό ερώτημα όμω είναι είμαστε τώρα στις ε, αποφασιστικές διαπραγματεύσεις για τη νέα νομική βάση των συστημάτων ελέγχου, των διευθυντικών ταμείων, του γεωργικού ταμείου. Τι στοιχεία θα ήθελε να μας δώσει το ελεκτικό συνέδριο για να συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις μας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Αλφε Πίπα. Από πλευράς Άλντε, ο κύριος Μούλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει αρχίσει να γίνεται παράδοση, θα λέγαμε, για το ελεγκτικό συνέδριο να παρουσιάζει τα στοιχεία του. Για μένα δεν αποτελεί αυτό έκπληξη. Είναι η 18η φορά που η ετοιμιγορία είναι αρνητική. Και κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Η Επιτροπή δείχνει μια σχετική αυταρέσκεια θα λέγαμε, γιατί η κατάσταση θα σταθεροποιείται και αυτό αποτελεί ένα καλό σημάδι. Έχει δοθεί μια καινούργια εξήγηση, κάτι, κάτι δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Αυτό το 3,9% που θεωρείται ποσοστό λάθους, λάθους από το ελεκτικό συνέδριο, λάβετε υπόψη τις ε, διορθώσεις και φτάνουμε στο 2%. Και αυτό είναι η διεθνής νόρμα και αυτό είναι κάτι που θεωρείται ικανοποιητικό. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν το δικαστήριο, ε, το, με συγχωρείτε, το ελεκτικό συνέδριο συμφωνεί με αυτό το επιχείρημα. Εγώ δεν συμφωνώ. Η κατάσταση σε ό,τι με αφορά δεν είναι τόσο καλή. Έχω την εντύπωση ότι η τάση δεν είναι προς τη σταθεροποίηση, αλλά είναι προς την επιδείνωση. Ήταν 3,3 πριν από δύο χρόνια, 3,8 και τώρα φτάσαμε στο 3,9 ποσοστό λάθους. Έχω την εντύπωση ότι από όποια πλευρά και να το δούμε αυτό δεν αποτελεί βελτίωση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κοινοβούλιο. Ε, εγώ προσπαθώ Προσπαθήσαμε τα πάντα τα τελευταία χρόνια. Δεν βοήθησε όμως τίποτα. Ζητήσαμε στην τελευταία διαθεσμική συμφωνία να υποβάλλονται αιτήσιες εκθέσεις. Μόνο πέρσι έκανε κάτι η Επιτροπή και υπέβαλε, δημοσιοποίησε την αιτήσια έκθεση. Ήταν κάπως αργά, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ. Δεν μπορέσαμε όμως να τα μελετήσουμε γιατί μας δόθηκαν στο πρωτότυπο. Είναι πρόβλημα αυτό για μένα, γιατί μεταξύ των άλλων δεν κατέχω την τσεχική γλώσσα. Συνεπώς θα πρέπει ο έλεγχος να βελτιωθεί. Το πιο σημαντικό εδώ, την τελευταία χρονιά, και κανένας δεν το ανέφερε αυτό το θέμα, είναι ότι έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Τι θεωρεί το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ποια είναι τα, οι απτές ε, βελτιώσεις που περιμένουν από αυτό, γιατί το Κοινοβούλιο περίμενε πάρα πολύ χρόνο για να υπάρξει μια απλούστευση των διαδικασιών. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ακούγαμε μερικά σχόλια με αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι περιμένουμε από αυτό για το Κοινοβούλιο, ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το 80% των ε, κονδυλίων ε, των πόρων δαπανώνται στις χώρες μέλη και κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Η ευθύνη της δημοκρατίας έγκυται στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε οι χώρες μέλη να κάνουν μία δήλωση σε το κατάλληλο πολιτικό επίπεδο. Είτε μιλάμε για ομόσπονδο κράτο, ε, είτε ε, οτιδήποτε άλλο. Κάποιος όμως, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι τέσσερις χώρες μέλη το έχουν ήδη πράξει στο παρελθόν. Υπήρξε ένα σημαντικό σημείο γι' αυτό το Κοινοβούλιο. Και πραγματικά θελήσαμε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος έγινε καταρχάς δεκτός για πρώτη φορά από τις χώρες μέλη. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερο αν το ελεγκτικό συνέδριο ανέλυε την απόδοση αυτών των τεσσάρων χωρών μελών που υπέβαλαν μια ετήσια δήλωση. Αν έλεγαν ότι η απόδοση είναι καλύτερη, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο σε σύγκριση με τον άλλο μελών, ποια είναι η άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου. Μήπως θεωρεί ότι δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι πουδενή ικανοποιημένο με τα αποτελέσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και ενώ ώψη των επόμενων εκλογών που θα είναι σε 1,5 χρόνο, έχουμε ακόμα ένα χρόνο μπροστά μας, την τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές. Πώς θα μπορούσαμε εμείς ως Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουμε ότι κάθε χρόνο θα μπορούσαμε να απαλλάσσουμε την Επιτροπή, ενώ 18 ολόκληρα χρόνια η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου υπήρξε ανητική. Σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε ως Κοινοβούλιο να χορηγούμε απαλλαγή όταν τα αποτελέσματα συνεχίζουν να είναι αρνητικά. Ευχαριστώ, ε, ο κύριος Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αν και δεν μπόρεσα να διαβάσω το σύνολο της έκθεσης. Από πρώτης απόψεως όμως φαίνεται να είναι πολύ πλήρης. Και έχει και παιδαγωγική θα έλεγα αξία με τις πίνακες που παραθέτεται. Κύριε Καντέρα, έχετε έρθει πολλές φορές να μας μιλήσετε, να μας παρουσιάζετε την ετήσια έκθεση και τα ίδια ακούμε κάθε φορά, σχεδόν τον ίδιο λόγο. Δεν φταίτε εσείς βέβαια γι' αυτό, αντίθετα. Πάντως με εκνευρίζει αυτή η κατάσταση. Δεν βλέπουμε να βελτιώνεται τίποτα. Και το σημαντικότερο, το πιο αρνητικό είναι ότι πρόκειται για το πρώτο δημοσιονομικό έτος όπου η δεύτερη επιτροπή Μπαρόσο έχει πλήρη ευθύνη. Πριν από ένα χρόνο θα μπορούσε να πει ότι ναι, είμαστε και εμεί τμήμα του προπολογισμού, αλλά δεν ήταν οι ίδιοι επίτροποι όλοι κτλ. Τώρα όμως είναι η πρώτη φορά που ο προϋπολογισμός τίθεται πλήρως στην ευθύνη της Επιτροπής Μπαρόσο 2. Κύριε Σεμέτα, έχουμε καλές σχέσεις έρχεστε εσείς συχνά στην Επιτροπή μας, αλλά ο λόγος που μας βγάλατε σήμερα αναρωτιέμαι με βάση αυτόν αν εσείς και οι συνάδελφοί σας είτε στον ίδιο κόσμο με μας ή στον πραγματικό κόσμο. Έχω μερικές αμφιβολίες. Οι αριθμοί που παίρνω εγώ από το ελεγκτικό συνέδριο δεν λένε, όπως είπατε εσείς, ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Το 2006 υπήρχε το περιθώριο λάθους 7,3 μετά μειώθηκε στο 3,3 όντως αλλά δεν βελτιώθηκε περαιτέρω τώρα έχουμε 3,9 από το 9 μέχρι σήμερα όμως αυξήθηκε κατά μισό της εκατό το περιθώριο λάθος δεν είναι και τόσο καλό αυτό ούτε πρόοδος και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου διαβάζω ότι οι τομεί πολιτικής όπου είχε, υπήρχαν τα περισσότερα λάθη ήταν η αλληλεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η ενέργεια, η απασχόληση, η ανάπτυξη και η έρευνα. Αυτά είναι σχεδόν όλος ο προϋπολογισμός. Και σε δύο μόνο τομείς, το είπαν και άλλοι αυτό, υπήρξε βελτίωση με λιγότερο ποσοστό λάθους δηλαδή γεωργία 2,3 και ανάπτυξη της υπαίθρου, ναι σημαντικά είναι, αλλά και στην ανάπτυξη 1,4 για την Επιτροπή μιλάω, για την Κομισιόν. Αλλά γενικά είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά λαθρό, όπως στις μεταφορές 6%. Συμφωνώ με τον κύριο Μολτέρ Υπάρχει η ευθύνη των χωρών μελών, το είπατε και εσείς κύριε Σεμέτα και είναι φανερό και από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Η περιφερειακή πολιτική, στην περιφερειακή πολιτική 60% των λαθών θα έπρεπε να είχαν ταυτιστεί από τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό ίσχυε και για πέρυσι, ούτε εκεί έγινε πρόοδος. Στη συνεργασία μας με τους διάφορους ηγητές λοιπόν είδαμε φέτος όπως είπε και ο κύριος Μολτερ, ότι πρέπει να βρούμε μια άλλη μέθοδο. Το Κοινοβούλιο προσπάθησε ήδη από μερικά χρόνια πριν να αναγκάσει να πείσει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν το πετύχαμε. Αυτός πρέπει να είναι ο κύριος στόχος ως προς την απαλλαγή. Δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς δεν ψέχουμε μόνο την Κομισιόν, ξέρουμε ότι και τα κράτη-μέλη, ότι τα κράτη-μέλη κάνουν τα λάθη. Αλλά αυτό πρέπει να είναι ο στόχος σας και ο δικός μας. Και για αυτή την απαλλαγή πρέπει να αναρωτηθούν οι επίτροποι, να ρωτήσουμε τους επιτρόπους να μας πούν με συγκεκριμένο τρόπο ρητά πώς σκοπεύουν να μειώσουν αυτά τα περιθώρια λάθους. Να τεθεί κάποιο χρονικό όριο κάποια προθεσμία. Και μετά πρέπει και προς το Συμβούλιο να δηλώσουμε στην τωρινή Προεδρία όταν θα έρθει να μας δει σε μερικές εβδομάδες και θα συζητηθεί η απαλλαγή για πρώτη φορά να μας δώσουν να μας πούν ακριβώς τι σκοπεύουν να κάνουν, να το κάνουν σοβαρά. Γιατί και αυτοί λένε κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν τα παίρνουν στα σοβαρά αυτά τα πράγματα. Και το Συμβούλιο ποτέ δεν είδε σοβαρά το θέμα της απαλλαγής. Το θεωρούν ένα τυπικό στοιχείο στην ενωσιακή ζωή, αλλά δεν είναι. Πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι ευθύνε των κρατών μελών, δηλαδή του Συμβουλίου. Τις αναφέρει το ελεκτικό συνέδριο. Αυτά τα δύο πρέπει να πούμε, να ζητήσουμε από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου να έρθει να μας μιλήσει αληθινά. Όχι απλώς ε, έτοιμα λόγια κάθε χρόνο τα ίδια. Σταματάω εδώ γιατί δεν μπόρεσα να διαβάσω την πλήρη έκθεση από χθες το βράδυ. Αντίθετα, γιατί αντίθετα από ό,τι μου είχαν υποσχεθεί δεν τη βρήκα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Θα την κοιτάξω όμως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, αριστερά. Σόρεν Σαντεγκάρτ. Σόρεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση που υπέβαλε. Θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα, αλλά θα ήθελα να κάνω και μερικά γενικά σχόλια. Το πρώτο ερώτημα αφορά την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από το πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου που αφορούσε τις δαπάνες. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο για να το βλέπει κανεί αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα το το αποκαλεί σφάλμα. Γιατί πραγματικά θα ήθελα, αν θα μπορούσατε να μου δώσετε μία ιδέα του πόσε δηλώσει κόστους έχουν γίνει. Γιατί όταν μιλάμε για πραγματικό σφάλμα, Αυτό σημαίνει ότι γίνονται υπερβολικές ε, δηλώσεις, ενώ μερικές φορές γίνονται λιγότερες δηλώσεις. Εάν συστηματικά δηλώνονται παραπάνω ποσά, αυτό σημαίνει ότι κινούμεθα σε ένα διαφορετικό τομέα. Δηλαδή, εσκεμμένα προσπαθεί κανείς να αποσπάσει περισσότερα χρήματα από όσα δικαιούται. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση που έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Έχουμε ένα παράτημα στην ηλεκτρονική έκδοση και με βάση αυτή την έκδοση διαπιστώσαμε ότι το αναμενόμενο περιθώριο στα σφάλματα πληρωνών πέρασε από το 3,4% στο 5,1%. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιο σχόλιο σε ό,τι αφορά την επίπτωση που έχει αυτό σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Ανάπτυξης. Η τρίτη μου ερώτηση αφορά το θέμα της ε, γεωργίας. Ως προς τη γεωργία παρατηρήσαμε μια σημαντική αύξηση στο σφάλμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου και παρακαλώ να τις επιβεβαιώσετε, έχουμε δει περιπτώσεις όπως στη Γεωργία και ιδιαίτερα στο 2011 να διεξάγονται περισσότερες έρευνες, περισσότεροι έλεγχοι. Εάν όντως ισχύει αυτό, αυτό, πέστε μου αν αυξηθεί ο αριθμός των ελέγχων, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του ποσοστού λάθους. Θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε δύο λόγια σε ό,τι αφορά τη σχέση με την αύξηση του εντοπιζόμενου αριθμού λαθών και των ελέγχων. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό ισχύει και για τους άλλους τομείς. Αύξηση λοιπόν του αριθμού των ελέγχων που γίνονται σε άλλες περιοχές και να δούμε κατά πόσον αυτό θα οδηγήσει στον εντοπισμό υψηλότερου ποσοστού λάθους. Τώρα, μία ε, παρατήρηση γενικότερη φύσης. Μεταξύ του 2006 και του 2009 είδαμε μία μείωση στο ποσοστό σφάλματος. Ακούσαμε, η Επιτροπή είπε ότι ε, σε εκείνη οφείλεται και αυτό έγινε μετά από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να το αναγνωρίσω αυτό, εάν οφείλεται η αναγνώριση αλλά το 2010 παρατηρήθηκε μια αυξητική τάση. Κινηθήκαμε προς την αντίθετη κατεύθυνση και η Επιτροπή είπε ότι αυτό ήταν μια σύμπτωση. Αφορούσε μια και μοναδική χρονιά και δεν θα μπορούσε να ε, αποδοθεί κάπου. Το 2011 είδαμε μια κίνηση προς την αρνητική κατεύθυνση. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι κατά πόσον είναι θέμα σύμπτωσης ή είναι θέμα που αφορά πολλού παράγοντε ε, Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη γι' αυτό, όπως ήταν υπεύθυνη και για όταν πηγαίναν καλά τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος Μόλτερ, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι αποφασιστική. Δεν μπορώ να φανταστώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάει στους ψηφοφόρους ενώ έχει παρακολουθήσει τα πράγματα να επιδεινώνονται διαρκώς σε διάστημα τριών ετών. Εάν δεν υπάρξει μία βελτίωση την επόμενη χρονιά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μία συγκεκριμένη κατάσταση. Ε, τα τελευταία 18 χρόνια οι λογαριασμοί της Επιτροπής απορρίπτονται από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό, γιατί εάν αποταθούμε στους ψηφοφόρους και εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους ότι για τρία συναπτά έτη υπήρξε πρόβλημα με τους λογαριασμούς και εκείνοι θα μας πούνε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και μετά η κυρία Ανδρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να φανταστώ τη θέση του Επιτρόπου γιατί ο προκάτοχός του ήταν υπεύθυνο και τον έλεγχο του προπολογισμού. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά, μία φορά το χρόνο, ε, υπήρχε αυτή η ανησυχία της αντιμετώπισης από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εργαζόμουν ε, ε, για εκείνο και εκείνη την εποχή όταν μιλούσαμε για αύξηση στο ποσοστού λάθους φαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των δεσμεύσεων και των πληρωμών για μία ακόμα φορά αυξήθηκε. Η Επιτροπή Προπολογισμού του Κοινοβουλίου θα επιθυμούσε περισσότερη περισσότερους πόρους ε, περισσότερη εξουσία και στην ουσία ε, αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις και δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε μετά. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς υπήρχε ένα πλεόνας με 1,5 δισεκατομμύρια. Το 2010 ήταν 20 ε, δισεκατομμύρια. Βλέπετε ότι δεν λείπουν τα χρήματα. Τα χρήματα έχουμε. Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί προσπαθούμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό αφού δεν είμαστε σε θέση να τα ξοδέψουμε όπω πρέπει. Αν κοιτάξουμε το περιθώριο σφάλματο στην έκθεση για 18η φορά δεν θα εγκριθεί. Αν κοιτάξετε το ποσοστό σφάλματος στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και της γεωργικής ανάπτυξης, θα δείτε ότι είναι υψηλό. Αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την Επιτροπή. και αυτό μας βοηθάει να φτάσουμε το 2-5% για, τις, ε, ε, για την ενέργεια και τις μεταφορές. Ενδεχομένως οι προσδοκίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες γιατί αυτή είναι μια πολιτική που αφορά τη γραφειοκρατία. Όταν υπάρχει γραφειοκρατία, όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί σε επίπεδο βρυξέλλων τι θα συμβεί σε κάθε μέρος της χώρας. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σκαρίφημα. Από τις Βρυξέλλες προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τι θα συμβεί στις χώρες μέλη από ένα κεντρικό επίπεδο και ενδεχομένω έχουμε φτάσει στα όρια του εφικτού. Ίσως θα μπορούσα να θέσω ένα ερώτημα εδώ. Όταν ε, μιλάμε για την ε, ενίσχυση στην ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάσκεψης έχει ένα περιθώριο σπάνιτος 5%. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι θα μπορούσατε να πείτε σε ό,τι αφορά το προπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη χρησιμοποιεί ε, την ενίσχυση του προπολογισμού για χώρε που δεν έχουν εμπειρία στον τομέα της καλής διακυβέρνησης. Στην ΑΕΤ, για παράδειγμα, ε, τα χρήματα δαπανώνται σωστά ή ελέγχεται μόνο το κατά πόσον έχουν σταλεί τα ποσά αυτά. Εσείς τι κοιτάτε μόνο, να έχουν εφαρμοστεί σωστά ε, τα προγράμματα και αν έχουν επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. κύριε Κυρία Αντρίεσεν, θα ήθελα να σας πω σε τι πλαίσιο συζητάμε την ετήσια αυτή έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Διανύουμε μια περίοδο κρίσης. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ζητούν μια αύξηση 7% για τον προπολογισμό του 2013. Ζητούν επίσης, ζητάμε εμείς μια αύξηση 5% για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συζητήσαμε το ποσοστό σφάλματος. Κοιτά όμως εδώ τη συχνότητα σφάλματος και είναι ανησυχητικό το να διαπιπτωσώσει κανείς το 50% των συναλλαγών για το μεγαλύτερο μέρος του προπολογισμού παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σφάλματος, πάνω από 50%. αναφέρθηκε ότι οι χώρες μέλη είναι υπεύθυνε γι' αυτό. Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη, γιατί η Επιτροπή έχει την εξουσία να βάλει τέλος στις πληρωμές όταν βλέπει ότι υπάρχουν ατασταλίες, ότι υπάρχουν ατυπίες. Οι φορολογούμενοι δίνουν τα χρήματά τους στην Επιτροπή και η Επιτροπή είναι εκείνη που έχει στα χέρια της την εξουσία για να δώσει ή για να σταματήσει τη χρηματοδότηση όταν θεωρεί ότι δεν χρησιμοποιείται σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω στον κύριο, τον κύριο Καλδέρα στην αναθεώρηση των συναλλαγών εντόπισε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή διέκοψε τις πληρωμές όταν διαπίστωσε ότι υπάρχουν ε, Πολλά υπόθηκαν σχετικά με το ότι το σφάλμα δεν είναι απάτη. Για μένα η δήλωση μη επιλέξιμο δαπανών ισούται με απάτη. Και στις χώρες μέλη αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη φυλακή κάποιον που θεωρείται υπεύθυνο. Θα μπορούσαν οι ελεκτέ να μου πούν αν αυτή είναι η άποψή του, εάν πιστεύουν ότι η έννοια του, του σφάλματο δεν ταυτίζεται με την έννοια τη απάτη. Αναφέρθηκε εδώ ότι η δήλωση των χωρών μελών θα ήταν μία λύση. Διαφωνώ και με αυτό. Οι χώρες μέλη στο σύνολό τους δεν μπορούν να αναλάβουν ευθύνη για δαπάνες ε, που τις διαχειρίζονται άλλοι φορείς στη χώρα. Πιστεύω ότι η λύση θα ήταν για μία φορά αυτό το Κοινοβούλιο να αρνηθεί την απαλλαγή προς την Επιτροπή. Τέλος, ο κύριος Καλντέρα αναφέρθηκε σε δίκαιους λογαριασμούς. Εγώ θα ήθελα να έχω κάποια διασφάλιση ότι είναι δίκαιη, γιατί στο τέλος του 2011 ο υπεύθυνος Επίτροπος για τον Προπολογισμό μας είπε το Φεβρουάριο ότι υπήρξαν, υπήρξε ένα έλλειμμα στο προπολογισμό, ενώ τον Απρίλιο υπήρξε πλεόνασμα. Εγώ δεν έχω εμπειρία σε οποιαδήποτε οργάνωση όπου η διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος του προπολισμού, μεταξύ του ελλείμματος και του πλεονάσματος ήταν τόσο μεγάλη σε διάστημα δύο μηνών. Θα ήθελα να πω ότι στην τελευταία έκθεση γίνεται αναφορά στην προχρηματοδότηση. Αυτή τη χρονιά δεν γίνεται, δεν κάνετε καμία αναφορά στην προχρηματοδότηση. Μπορείτε το σχολιάσετε κύριε Καλντέιρα. Ευχαριστώ κυρία Αντρέασεν. Τα ερωτήματα γίνονται όλο και περισσότερα. Έχω άλλους δύο που θέλουν το λόγο πριν παρακαλέσουν να δώσουν απαντήσεις. Η συνάδελφος Ίνια Κρέσλε. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η φετινή έκθεση. Όπως είπε και ο συνάδελφος Μπίμπερ, είναι πιο διαφανής από τον προηγούμενο. Θέλω να θυμηθώ πώς ήταν η κατάσταση ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου πέρυσι. Νομίζω ότι κάθε χρόνο το συνέδριο αλλάζει τα κριτήριά του, τον τρόπο συλλογής στοιχείων. Ε, πολλές φορές η συνδιαχείριση με την απευθείας διαχείριση, οπότε δεν είναι σαφής η κατάσταση. Μας δημιουργεί πολλές ε, ανησυχίες. Αν δούμε τι αλλάζει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, δεν ευνοείται έτσι η διαφάνεια αν αλλάζουμε τι δαπάνες ε, λαμβάνουμε υπόψη κατά διάρκεια του χρόνου. Για τα διαρθρωτικά ταμεία και την ενέργεια περιφερειακή και μεταφορές. Και εδώ ε, μπερδεύουμε τους ε, τρόπους διαχείρισης, άρα δεν υπάρχει διαφάνεια. Θα ήθελα να δω λοιπόν πώ ε, διανέμονται αυτά και για την ε, ανάπτυξη και εσωτερικέ πολιτικέ. Το ίδιο διαπιστώνουμε. Και για τη συνοχή τη διαπιστώνω υπήρξε επιδείνωση τη κατάσταση. Δεν αναφέρεται σαφώ αυτό στην έκθεση όσο θα έπρεπε. Ούτε μία στι πέντε πληρωμέ δεν είναι χωρί σφάλματα. Δηλαδή, τέσσερι από τι πέντε έχουν σφάλματα. Πέρυσι ήταν 75%. Τώρα πλησιάζει το 80% το ποσοστό πληρωμών όπου υπάρχουν σφάλματα. Πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Τι γίνεται με τη συνοχή. Τι γίνεται με τη διαχείριση της συνοχής στα κράτη-μέλη. Γιατί εδώ έχουμε τα προβλήματα στις εθνικές διοικήσεις. Πρώτο λοιπόν αυτό, να μας πείτε τι γίνεται το Ταμείο Συνοχής. Και για το θέμα αυτής της σύγχυσης ε, που προανέφερα. Τρίτο, έχουμε χώρες όπου έχουμε συγχρηματοδότηση 100% δηλαδή, όχι συγχρηματοδότηση, χρηματοδότηση 100% από την ε, Ένωση. Πώς το βλέπει αυτό το συνέδριο. Τέτοια ποσοστά δεν είχαν ποτέ. Τι πορίσματα εξάγεται από αυτή την κατάσταση. Οι χώρες οι οποίες παίρνουν 100% γιατί δεν μπορούν να δαπανίσουν ούτε καν μια πλήρη κοινοτική χρηματοδότηση. Θα ήθελα επίσης παρακαλώ να μας πείτε για, τον, ε, για την ποιότητα των εξωτερικών ελέγχων. Διότι με ανησύχησε το ότι είδα ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν και αυτοί υψηλό ποσοστό σφάλματος. Πάνω από τους μισούς. ελέγξατε το 25% και το 14% είχε σφάλματα. Πάνω από το μισό δηλαδή. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορούμε ούτε καν ε, σε αυτούς που υποτίθεται είναι οι δήμονες να έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτούς που επιφορτίζουν τα κράτη-μέλη για να κάνουν εξωτερικούς ελέγχους και η Επιτροπή. Αν δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τέτοιους ελέγχους δεν ξέρω πού μπορούμε να βασιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τελευταίος ο συνάδελφος Μπαλζίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι άλλοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεσή του. Καλό θα ήταν βέβαια να είχαμε λάβει το κείμενο λίγο νωρίτερα για να καταλάβουμε ευκολότερα πού ακριβώς υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε έτσι πρόχειρα. Το ερώτημά μου προς τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου είναι το εξής. Κοιτάζοντας τα στοιχεία που δίνετε και σε αυτήν και σε προηγούμενες εκθέσεις σας, πόσο αξιόπιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι. Από το 98 η Κομισιόν μας λέει ότι δεν έχει αξιόπιστα στοιχεία από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό δεν μπορεί να θεωρείται υπόλογη και υπεύθυνη για τα στοιχεία που χορηγεί στο συνέδριο. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν να δώσουν τα στοιχεία που αφορούν τις απάτες. Και άλλος το είπε αυτό. Όταν μιλάμε για τον ορισμό του περιθωρίου λάθους υπάρχει μια διαφορά μεταξύ λάθους και απάτης. Δηλαδή αναγνωρισμένης απάτης. Πρέπει να αρχίσουμε να αναλύουμε κάποτε τις γενικές αρχές εφαρμογής του ενωσιακού προϋπολογισμού στις τωρινές δημοσιονομικές προοπτικές στις επόμενες. Όταν μπήκαμε στην Ένωση, αυτό που κυρίως θέλαμε ήταν να απαλλαγούμε επιτέλους από τις ελλείψεις που είχε η δημόσια διοίκηση στις χώρες μας με βάση τα ενωσιακά χρήματα. Αλλά η στήριξη της Ένωσης φτάνει μόνο στο 5 με 10% του εθνικού προϋπολογισμού και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να στοχευθεί καλύτερα αυτή η δημοσιονομική στήριξη της Ένωσης, η χρηματική στήριξη. Η ετήσια έκθεση που συζητούμε σήμερα συμπεριλαμβάνει μια δήλωση ότι, δηλαδή, σε σύγκριση με το 10, ο το περιθώριο λάθους έχει αυξηθεί από τα 400 εκατομμύρια σε ένα δισεκατομμύριο. Τεράστιο ποσό που δείχνει δύο δις. Αυτό είναι τεράστιο ποσό και δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει πιο συγκεντρωτικά να εξετάζουμε τις αρχές της εφαρμογής του ενωσιακού προϋπολογισμού. Βλέπουμε ότι συχνά μετά από εκλογές στα κράτη-μέλη εμφανίζονται καινούργοι υπεύθυνοι ορισμένων τομέων που δεν είναι έτοιμοι δεν καταλαβαίνουν ακόμη εύκολα τους πολύπλοκους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν. Άρα ήδη από τώρα πρέπει να συζητήσουμε τις βασικές αρχές της εφαρμογής, της χρήσης της ευρωπαϊκής στήριξης, να μας πει ιδέες η Κομισιόν για αυτό το θέμα και να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε τα προβλήματα που συζητάμε εδώ για 18η φορά. Ευχαριστώ. Οπότε τώρα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο Καλδέρα και τον Επίτροπο Σεμέτα να πάρουν το λόγο. Ποιος θα ήθελε να μιλήσει πρώτος, ποιο θα ήταν σκοπιμότερο. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι ευγνώμων για τα σχόλια που προήρθαν από τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής και που αφορούν το έργο που επετέλεσαν στο ελεκτικό συνέδριο όσοι ασχολήθηκαν με αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Λαμβάνω υπόψη μου ότι σε μία περίπτωση μας επιφυλάξατε ένα, ένα ευμενές ε, σχόλιο ότι είμαστε διαφανείς, Σας σε μια άλλη περίπτωση δεν είπατε, είπατε ότι δεν είμαστε. Υπάρχει, είναι κάπως ναι, νεφελώδες αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει και μια σχετική αδιαφάνεια. Η συγκρισιμότητα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και βεβαίως Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και νομίζω ότι καταφέραμε να παρουσιάσουμε τις αλλαγές που επήλθαν με έναν τρόπο διαφανή, δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερο έλεγχο και δώσαμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή αυτή να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα που υφίστανται στην αρχική πολιτική και στον γεωργικό τομέα. Βεβαίως θα πρέπει να αποκαλύψουν τις αλλαγές, ποιες είναι οι ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις και τι θα γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή έχει στη διάθεσή της αυτές τις πληροφορίες και με απόλυτη διαφάνεια. Το γεγονό ότι οι πληρωμέ διαλύουν το πέμπτο έτο τη περίοδου προγραμματισμού βεβαίω έχουν ένα διαφορετικό προφίλ, αλλά τα συστήματα που βρίσκονται στην βάση αυτών των πληρωμών παραμένουν σταθερά. Συνεπώ. συμφωνώ ενδεχομένω με τον κύριο Στάσε, επαναλαμβάνομαι για πέμπτη ε, χρονιά. Ξανακοίταξα τι ομιλίε μου το Σαββατοκύριακο και πραγματικά διαπίστωσα ότι επαναλαμβάνομαι. Για πέμπτη συναπτή χρονιά λέω εξ ονόματο του ελεκτικού συνεδρίου ότι θα πρέπει να έχουμε πιο απλό, απλά προγράμματα με σαφή καθορισμό στόχων που μας επιτρέπουν εύκολα να ε, ελέγχουμε το αποτέλεσμα και να έχουμε σωστούς μηχανισμούς. Αυτό θα ήθελε το ηλεκτρικό συνέδριο και αυτό εκφράζεται στη σειρά από τομεακές προτάσεις που τώρα είναι υποσυζήτηση και που αφορούν τον τομέα της γεωργίας, ε, του Ταμείου Περιφερειακής Συνοχής και στην ουσία αυτό είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Και τονίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιβάλλουμε μηχανισμούς, ενισχυμένους μηχανισμούς και θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου κόστους ωφέλους στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μηχανισμών. Αυτά είναι και θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Κατά την άποψή μας, το νέο δημοσιονομικό κανονισμό διατυπώσαμε την άποψη ότι υπάρχει ένα δυναμικό. Εάν οι τομεακοί κανόνες ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στο δημοσιονομικό κανονισμό, ε, ε, στο κανονισμό, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν ορισμένες ε, δηλώσεις οι οποίες έχουν σχέση με τον κανονισμό αυτό, ακόμα και πριν να τεθεί σε εφαρμογή. Νομίζω ότι είναι καινοτομία το γεγονός ότι και το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξέφρασαν άποψη για αυτό το θέμα και το Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις και από την αρχή υπήρχε ανάγκη να δοθούν ορισμένες διευκρινήσεις ως προς κάτι που δεν είχε εφαρμοστεί. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και πιστεύω ότι για λόγους απλούστευσης στον ε, τομέα των, κρατικών προ, ε, των δημοσίων συμβάσεων υπάρχει μία ε, γνωμοδότηση το 2011 και μία συζήτηση για το πώς θα μπορούσαν να απλοποιηθούν οι δημόσιες συμβάσεις και κατεβλήθη όντως μία προσπάθεια να γίνει απλοποίηση, παράλληλα όμως με το σεβασμό των βασικών αρχών της ενιαίας αγοράς. Ο κύριος Μούλτερ τόνισε, αναφέρθηκε σε αυτό που θα μπορούσαμε να αναμένουμε από το νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Ακούστε, θα πρέπει να δούμε τι συμφωνία, τι εφαρμογή θα υπάρχει των τομεακών κανονισμών. Πρέπει να περιμένουμε. Είπατε επίσης ότι εάν δούμε τις διορθώσεις και τις αφαιρέσουμε από το ποσοστό λάθους, θα μπορέσουμε να βρούμε το πραγματικό ποσοστό λάθους. Εγώ θα πρόσεχα στο σημείο αυτό. Γιατί οι δημοσιονομικές διορθώσεις συνδέονται με πληρωμές που έγιναν το παρελθόν, όχι το 2011. Εγώ θα ήμουν υπέρ του να υπάρξει αυτή η μεθόδευση εάν οι διορθώσεις αφορούσαν πληρωμές αυτής της χρονιάς. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, αφορούν προηγούμενες χρονιές και όλοι οι μηχανισμοί διορθώσεων αφορούν διορθώσεις των προηγούμενων ετών, όχι του 2011. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πιστεύουμε ότι το γεγονός ότι απεκάλυψε η Επιτροπή αυτές τις πληροφορίες σηματοδοτεί μια μεγάλη πρόοδο και αν κοιτάξουμε την έκθεση θα διαπιστώσουμε ότι οι επιφυλάξεις από τις γενικές διευθύνσεις αφορούσαν το σημείο τα σημεία που υπήρχαν τα προβλήματα. Συνεπώς έχουμε αυτές τις πληροφορίες, υπάρχουν, είναι διαφανείς και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές και να αναπτύξουμε στο μέλλον της δράσης μας. Το ερώτημα του πού οφείλονται τα πολλαπλά λάθη στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης που, είναι το, που βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Πιστεύω ότι η εξήγηση βρίσκεται στην έκθεση που υποβάλαμε. Τα συστήματα που βρίσκονται στη βάση των πληρωμών στο συγκεκριμένο αυτό τομέα δεν εφαρμόζονται πλήρως. Συνεπώς δεν μπορούν να προλάβουν και να ανοιχνεύσουν τα λάθη. Εγώ παρέθεσα το παράδειγμα της αποτυχίας του πρώτου επίπεδου ελέγχου που δεν εφαρμόθηκε από τον οργανισμό πληρωμών όταν έλεγχε τα προγράμματα που αφορούσαν την αγροτική ανάπτυξη. Βεβαίως αυτό συνδέεται και με την αποτυχία της πρώτης γραμμής άμυνας ε, που ε, χρησιμοποιούν οι χώρες μέλη και που αφορά τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ε, Ένωσης. Βεβαίως μετράνε και οι κανόνες των χωρών μελών, γιατί έχουμε καθορίσει ένα σύστημα που βασίζεται στην επιλεξιμότητα. Αυτές οι συνθήκες όμως επιλεξιμότητας δεν συνδέονται, ε, δεν ε, τίθεται σε επίπεδο κοινότητας, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών. Κάθε χώρα έχει τις δικές της συνθήκες επιλεξιμότητας. Και από αυτό προκύπτει ε, ε, καθιστά τα πράγματα πολύπλοκα. Ενώ εμείς βρισκόμαστε σε αναζήτηση απλούστευσης. Ενώ κοινά, στο κοινό ε, κανονισμό βλέπουμε ότι υπάρχουν έξι επίπεδα νομοθεσίας. Συνεπώς η απλούστευση εξαρτάται και από εμά και από το Συμβούλιο και από τις χώρες μέλη που κάποια στιγμή θα καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και θα κάνουν τις σωστές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Με χαρά θα απαντούσα γραπτός στα αξιότιμα μέλη, σε πολλά από τα αξιότιμα μέλη. Ένα άλλο ε, θέμα που θίξατε Περισσότερο έλεγχο συνεπάγεται περισσότερα λάθη, ταυτίζεται με την έννοια των περισσότερων λαθών. Δεν ξέρω ποια είναι η βάση για αυτό που λέτε θα μπορούσατε να πείτε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ελέγχων και σφαλμάτων και διαπίστωση σφαλμάτων. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, τα περισσότερα σφάλματα δεν προκύπτουν από τους περισσότερους ε, ελέγχους. Νομίζω ότι εάν γινόντουσαν περισσότεροι έλεγχοι δεν θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση του να προσπαθούμε τον υστέρο να τα διορθώσουμε τα πράγματα. Ας πούμε, ε, οι δασόδεις ε, εκτάσεις. Αν ας πούμε δεν επικαιροποιούνται τα στοιχεία, ε, εάν δεν εντοπίζονται οι περιοχές που βρίσκονται δάση, η το αίτημα αυτό υποβάλλεται και καταβάλλονται τα, τα κονδύλια, τα, τα, τα ποσά. Και ενδεχομένως μετά από 20 χρόνια γίνεται μία άλλη επικαιροποίηση. Υπάρχουν όμως τα στοιχεία. Θα πρέπει να καταβληθεί μία προσπάθεια από τις χώρες μέλη για να α, δίνεται σε επικαιροποίηση ας πούμε των βοσκότοπο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το γεγονός ότι οι εθνικοί οργανισμοί πληρωμής ελέγχουν και υπάρχει ένα κτίριο το οποίο δεν προσφέρεται, δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση και χρηματοδοτείται, αποδεικνύει ότι υπάρχει μια δυναμία στο σύστημα ελέγχου. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά σφάλματος στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης φέτος. Τα συστήματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε και ακόμα και αν διεξάγονται έλεγχοι, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν λάθη. Περισσότεροι έλεγχοι δεν συνεπάγονται και περισσότερα σφάλματα. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Ταμείο Ανάπτυξης. Αναφέρθηκε λοιπόν το θέμα του Ταμείου Ανάπτυξης. Υπάρχουν λόγοι στους οποίους ε, οφείλεται η αύξηση του ποσοστού λάθους. Τα συστήματα είναι βεβαίως της αρμοδιότητας ε, του Γενικού Διευθυντή. Θα μπορούσαμε βεβαίως ε, να παραθέσουμε και επιτοπίως παραδείγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που πήγαν άτομα και διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σχετικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν στο δείγμα σας σε ένα συγκεκριμένο έτος υπάρχουν σφάλματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις, ενδεχομένως και το ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Αυτός είναι ένας τομέας που πιστεύουμε ότι η θέση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ε, ξεκάθαρη. Σας απασχολεί το θέμα του λάθους. Βεβαίως ε, παρατηρήσαμε ότι αυξήθηκε η συχνότητα από πέρσι σε φέτος σε ορισμένες ε, περιοχές σε σύγκριση με άλλες. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για συχνότητα σφαλμάτων είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι ακριβώς ε, εννοούμε. Να μην ε, υπάρχει σύγχυση με άλλους τομείς. Η συχνότητα σφαλμάτων είναι ένα μέτρο των ε, προβλημάτων σε ένα πληθυσμό που ελέγξαμε. Σε ορισμένες ε, περιπτώσεις η επίπτωση είναι μεγάλη, σε άλλη περίπτωση δεν είναι μεγάλη αν μιλάμε για σφάλματα. Αν ας πούμε είμαστε στην, στον τομέα της βιομηχανικής ε, αλήσου που παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας, αυτό σημαίνει ότι το τάδε αυτοκίνητο ε, κάθε 44ο αυτοκίνητο παρουσιάζει προβλήματα. Δεν σημαίνει όμως ότι και τα 44 αυτοκίνητα έχουν προβληματικό κινητήρα ή έχουν ένα καθρέφτη που δεν είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση. Αυτό, αυτό είναι η συχνότητα. Όταν ε, μιλάμε για το πιθανότερο λάθος, ε, μιλάμε για την ε, επίπτωση που έχουν αυτά τα λάθη, πώς επηρεάζουν οικονομικά τον προϋπολογισμό. Και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τα τελευταία τρία χρόνια και υπάρχουν βεβαίως ορισμένες ε, διακιμάσεις πάντοτε υπάρχουν διακοιμάσεις, γιατί δεν είναι πάντοτε σταθερός ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός είναι ένα δείγμα όταν μιλάμε για πληρωμές. Υπάρχουν λοιπόν διακοιμάσεις και αυτό το είδος των διακοιμάσεων πάντοτε παρατηρούνται. Αλλά τα τελευταία τρία χρόνια το διάστημα ε, των ε, συμβαλμάτων αυτών είναι σχετικά σταθερό. Δεν είναι όμως τέτοιο που να μπορούμε να πούμε ότι αν αφαιρέσουμε αυτές τις διορθώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ε, θα φτάσουμε στο 2%. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι, δεν, δεν είναι θεμητό το να θεωρούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν στοιχεία ότι η Επιτροπή διέκοψε τις πληρωμές και ε, έκανε διορθώσεις εκεί που εντοπίστηκαν ατασταλίες. Υπάρχουν παραδείγματα περιπτώσεων που η Επιτροπή μάζεψε και πάλι, πήρε πάλι πίσω, τα συγκέντρωσε τα ε, ποσά που είχαν εντοπιστεί από το ελεκτικό συνέδριο. Υπάρχουν περιπτώσεις και το, στο κοινωνικό ταμείο και σε ό,τι αφορά την πολιτική ε, έρευνας τις επενδύσεις ποσών τα οποία ε, απέσυρε η Επιτροπή. Δύο λόγια για, την, ε, για τις τελευταίες ερωτήσεις από την κυρία Κρέσλερ. Θα ήθελα να αναφέρω γιατί η εξωτερική έλεγχη δεν είναι αξιόπιστη, γιατί δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στους εξωτερικούς ελεγκτές. Ιδιαίτερα στους τομείς όπου οι ελεγκτές έκαναν αυτή την έρευνα και δεν ε, στάθηκαν στο ύψος της αποστολής τους. Δηλαδή δεν ανείχνευσαν τα προβλήματα που εντόπισε μετά το ελεκτικό συνέδριο. Και αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα θα δείτε ότι θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις γιατί οι ελεκτέ δεν έδωσαν τι σωστέ πληροφορίε στην Επιτροπή. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη τη. Εμείς ε, εργαζόμαστε στον τομέα της διαδικασίας πιστοποίηση έτσι ώστε να έχουμε πιο αξιόπιστες πληροφορίες. Και πάλι όμως χρειαζόμαστε πιο αξιόπιστες πληροφορίες από τις χώρες μέλη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από αυτή την έκθεση. Και να θέσουμε περαιτέρω το ερώτημα στην Επιτροπή να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχουν εκθέσεις για, για τα αποτελέσματα να, και να γίνεται μία αναφορά στην αποτελεσματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξουν περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες. Και αυτό βεβαίως εξαρτάται και από τις πληροφορίες που θα παράσχουν οι χώρες μέλη που πρέπει να είναι αξιόπιστες. Τώρα η συχνότητα της συντοχής είναι υψηλή αλλά Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τον τομέα της συνοχής δεν θα πρέπει να συγχαίουμε με το Ταμείο Συνοχής. Ο τομέας ε, της ενέργειας και των μεταφορών κατελείπει το Περιφερειακό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής καθώς και ταμεία που αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη συνοχή, δεν μιλάμε για το Ταμείο Συνοχής αυτό καθ' αυτό. Μιλάμε για αυτούς τους τομείς περιφερειακής πολιτικής που αφορούν τις 27 χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένου εδώ και, το, εδώ και το Ταμείο Συνοχής. Και πάλι τα προβλήματα είναι παρεμφερή με τα προβλήματα ε, που αφορούν άλλους τομείς. Καταρχάς έχουμε μία καθυστέρηση στην αρχή γιατί γιατί μόλις γίνει μία συναλλαγή, μία αλλαγή, η Επιτροπή πιστο... έχει ε, ε, την επικοινωνία με τις αρχές και αυτό είναι καλό, γιατί αν παρατηρήσετε την τάση ακόμα στον τομέα της συνοχής, διαπιστώνετε ότι σε γενικές γραμμές συγκρίνεται το 7 με το 5,1. Και αν κοιτάξετε το κοινωνικό ταμείο, για πρώτη φορά υπάρχει μία ξεχωριστή αξιολόγηση, που είναι κάτι λογικό. Συνεπώς, αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις στις πληρωμές. Υπάρχουν εκρεμίσεις. Ε, δεσμεύσει στο, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, ταμείων, διαθετικών ταμείων και ταμείων συνοχή. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι τώρα οι χώρες μέλη ζητούν επιστροφές σε ψηλότερα επίπεδα και επικεντρώνονται ε, επικεντρώνουν αυτά τα αιτήματα, δημιουργεί προβλήματα ταμιακής ροής για την ε, Επιτροπή. Δεν θα πρέπει όμω να συγχαίρεται αυτό με τις προβλέψεις του προπολογισμού. Οι προβλέψεις του προπολογισμού είναι αυτό που είναι. ενδεχομένω. οι χώρες ε, μέλη κάνουν προβλέψει για τι ε, δαπάνες και δεν είναι οι ίδιες, αλλά οι λογαριασμοί ε, αντικατοπτρίζουν την τελική θέση και υπάρχουν βεβαίως οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί και τα μέλη το γνωρίζουν καλύτερα από μένα. Δεν θα συνέχεια λοιπόν τα δύο αυτά σημεία. Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι μακρηγόρησα πολλά από τα θέματα, δεν τα απάντησα και βεβαίως είμαι στη διάθεση των μελών να απαντήσω στα κρεμή ερωτήματα γραπτός. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Καλντέρα. Ξέρω ότι πρέπει σε λίγο να εγκαταλείψετε τη συνεδρίαση. Αναφέρομαι λοιπόν σε ένα από αυτά που είπατε, δηλαδή ότι το λεκτικό συνέδριο επί πολλά έτη τονίζει το γεγονός ότι πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός και να απλουστευτεί ώστε η Κομισιόν και πάνω από όλα τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν σαφώς ποιοι είναι οι στόχοι. Όπως έλεγε και ο Γκέτε, πρέπει ο άνθρωπος να συνεχίσει την προσπάθεια πέραν από το απλό περιθώριο λάθους για μας. προσπάθειά μας πρέπει να είναι να παίρνουμε μαθήματα από τα παθήματα. Εσείς εδώ και πολλά χρόνια στις εκθέσεις σας διατυπώνετε σχόλια που ακόμη ισχύουν. Όλοι βλέπουμε ότι γίνονται τα λάθη. Ανθρώπινο είναι αυτό. Δεν μπορεί ποτέ μια διοίκηση να μην σημειώσει κανένα λάθος. Αν όμως επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, ή δεν υπάρχει καμία πρόοδο σε ορισμένους τομείς, τότε πρέπει να ταυτίσουμε τις δυσκολίες, ιδίως εμείς οι πολιτικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για μας είναι πολύ σημαντικό εργαλείο η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί δεν μπορούμε να εξετάσουμε απευθείας μόνοι μας τη διοίκηση και είναι επίσης πολύτιμη η έκθεσή σας και για την Κομισιόν γιατί έχει διαφορετική προσέγγιση από τους δημοσιονομικούς ελέγχους της. Επίσης αναφερθήκατε στη μέθοδο που ακολουθείτε τους τυχαίους ελέγχους. Για μας πάντως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτή η μέθοδος ακολουθείται και εξ ονόματος της Επιτροπής μας θα ήθελα να πω πρώτον ότι η έκθεσή σας και η αιτήσια και οι ειδικέ είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά μας. και για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Πολλά από τα ερωτήματα που δεν απαντήσατε σήμερα θα ξαναεξεταστούν και κατά τη διαδικασία της απαλλαγής που σε λίγο θα αρχίσει και με ακροάσεις επιτρόπων στην Επιτροπή μας. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν κύριε Καλδέρα σας ευχαριστώ και προσωπικά αλλά και, όλοι, και όλους τους συναδέλφους σας στο ελεγκτικό συνέδριο. Ο κύριος Καλδέρα έχει και άλλες υποχρεώσεις βέβαια. Αυτό κατανοούμε όλοι και τώρα ζητώ από τον Επίτροπο Σίμητα να πάρει το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούσαν την Κομισιόν. Όχι για μεμονωμένους τομείς, αλλά γενικότερα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος απαντώντας στις ερωτήσεις. Δεν ήταν και τόσο πολλές που αφορούσαν άμεσα την Κομισιόν. Γενικά το θέμα που ετέθη περισσότερο ήταν πώς αξιολογούμε το περιθώριο λάθους που διαπιστώθηκε το 11. θα επαναλάβω ότι το 3,9% του λάθους δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Ιδίως αν σκεφτείτε ότι όλα τα προγράμματα ήδη λειτουργούν εδώ και αρκετό καιρό. Το 2009 το περιθώριο ήταν 3,3% αλλά αυτό αφορούσε τότε προκαταρκτικές πληρωμές και όχι τις λειτουργικές και τελικές και γι' αυτό υπάρχει περισσότερο περιθώριο λάθους. Τώρα όλα τα προγράμματα βρίσκονται στη φάση των ενδιαμέσων και τελικών πληρωμών και παρόλα αυτά το περιθώριο λάθους είναι κάτω του 4%. Επίσης άλλαξε η μεθοδολογία του ελεκτικού συνεδρίου και αυτό αύξησε κατά 0,1% το περιθώριο λάθους. Επίσης, ήδη φτάσαμε, μειώσαμε τα λάθη σε επίπεδο τέτοιο ώστε είναι πολύ πιο δύσκολο σήμερα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια να υπάρξει σημαντική βελτίωση. Κάποτε ε, το περιθώριο λάθους ήταν 7,3 ή 9% πρέπει να καταλάβετε ότι φτάνουμε σε όρια, στα όρια της δυνατής πρόοδου που μπορεί να γίνει στο περιθώριο λάθος. Οι διορθώσεις που μπορεί να γίνουν είναι θέμα που πρέπει να γνωρίζετε ότι γίνονται από την Κομισιόν σε πολυετή βάση, ενώ οι εκθέσεις του ελεγκτικού είναι ετήσιες. Και γι' αυτό το 11 έγιναν διορθώσεις της τάξης του 1,5% και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Συμφωνώ βέβαια με τον πρόεδρο Καλτέρα ότι είναι σημαντικό αυτό όταν κάνουμε την αξιολόγηση του 11 γιατί στο τέλος του πολυετούς πλαισίου θα ληφθούν τότε υπόψη αυτές οι διορθώσεις και τα εναπομένα λάθη και οι ανακτήσεις. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη σημαντική βελτίωση που σημειώθηκε στον τομέα της συνοχής από 7,7% σε 5,1% και μάλιστα στην ε, φάση πλήρους λειτουργίας του προγράμματος για τις δαπάνες, ιδιαίτερα στα κοινωνικά ταμεία όπου ήδη πλησιάζουμε στο επίπεδο λάθους που είναι το οριακό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω το γενικότερο σημαντικό θέμα του ότι μάλλον για πρώτη φορά η αξιολόγηση του περίπτωσης λάθους στις αιτήσιε εκθέσεις των γενικών μας διευθυντών ανταποκρίνονται πολύ στην ίδια την αξιολόγηση του συνεδρίου. Άρα τα συστήματα έχουν πράγματι βελτιωθεί ως προς την προετοιμασία των εκθέσεών τους και πρέπει να τονίσω ότι σε όλους τους τομείς όπου αυξήθηκαν τα περιθώρια λάθους όπως στην ανάπτυξη της υπαίθρου ή στην ε, έρευνα σε αυτούς τους τομείς έχουν γίνει παρατηρήσεις και, και από τους δικούς μας διευθυντές και ε, οι αρμόδιοι γενικοί διευθυντές έχουν ε, κάνει και προτάσεις και προτάσεις για βελτίωση με τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν. Και οι συνάδελφοί μου, οι άλλοι επίτροποι που θα έρθουν να σας μιλήσουν για τη γεωργία συγκεκριμένα, για τη συνοχή και για την έρευνα, θα σας τα αναφέρουν αυτά, τις λεπτομέρειες δηλαδή των προτάσεων που έκαναν οι γενικοί διευθυντές για την θεραπεία όλων αυτών των προβλημάτων. Όσο για το κατά πόσον προσέχουμε το θέμα της διακοπής πληρωμών, ναι, το προσέχουμε. Όταν διαπιστώσουμε, αν διαπιστώσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σε κάποιο κράτος μέλος, αμέσως διακόπτουμε τις πληρωμές και το 11, 91 τέτοιες διακοπές κάναμε σε ύψους 2,6 συνολικά δισεκατομμυρίων. Και φέτος αν και δεν έχει λήξει ακόμη το έτος, 89 διακοπές πληρωμών και 4 διακοπές. Και 4 πλήρες αναστολές. Βλέπετε λοιπόν πρόσφατο το καινούργιο αυτό σύστημα έχει ήδη αποτελέσματα. για το μέλλον συμφωνώ με τον κύριο Γκάγερ πρέπει να προσέξουμε περισσότερο το θέμα του επίπεδου λαθών που κάνουν τα κράτη-μέλη. Οι δύο συνομοθετικές αρχές συμφώνησαν επ' αυτού και αυτό είναι επίσης πρόοδος. Ο κύριος Μούλτερ ρώτησε ποια είναι τα ωφέλη του δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι σημαντικά. Έχουμε την ετήσια δήλωση διαχείριση την πολιτική δήλωση, αξιολόγηση του κόστους των ελέγχων και τους κινδύνους δημιουργίας λαθών κατά αυτούς. Νομίζω λοιπόν ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός είναι σοβαρή βελτίωση. Βέβαια δεν αρκεί, γιατί πρέπει αυτά που προβλέπει να εμφαίνονται να εφαρμόζονται και στην κατατομέα ανάλυση. Και το θέμα των όρων που βάζουμε στη νέα νομοθεσία δεν παραλείπονται ποτέ. Και συζητιέται ακόμη το θέμα και από τους δύο συνομοθέτες επίσης προτείναμε καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις, δηλαδή τα κράτη-μέλη που κάνουν λάθη, που έχει ταυτίσει το συνέδριο η δική μας έλεγχη, να οδηγούν σε μείωση της χρηματοδότησης που δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή από το υπάρχον σύστημα, από την υπάρχουσα νομοθεσία. Η πρόταση αυτή όμως αμφισβητείται από μερικές χώρες μέλη. Πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ζητάει και να πιέζει για την έγκριση των προτάσεων αυτών της Κομισιόν. Τέλος ευχαριστώ όλους εκείνους που έλαβαν το λόγο σήμερα. Όπως συνήθως η Κομισιόν θα σας δώσει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε για την καλύτερη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής και εγώ και οι συνάδελφοί μου επίτροποι θα έρθουν όποτε χρειαστεί για να συζητήσουμε κάθε κεφάλαιο λεπτομεριακά στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε Σίμητα και τώρα ο συνάδελφος Γκάγκερ για να καταλήξει ως εισηγητής. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά σχόλια. Ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο. Τα μέλη του συνεδρίου είναι μερικοί ακόμα εδώ, οι περισσότεροι όμως χρειάστηκε να φύγουν γιατί ο πρόεδρος Καλτέρα τώρα κάνει την συνέντευξη τύπου του για την παρουσίαση τη ετήσιας έκθεση Ευχαριστώ πάρα πολύ το συνέδριο, τα μέλη του συνεδρίου για την θαυμάσια συνεργασία που μας ε, υποβάλλει πολλές προτάσεις για τις περαιτέρω ενέργειές μας για καλύτερο δήμο, συνομικό έλεγχο των ε, κοινοτικών δαπανών. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Σεμέτα. Βεβαίως θα τα ξανασυζητήσουμε και σε άλλες συνθέσεις αυτά. Όπως ξέρετε, διάφοροι επίτροποι που φέρουν την κύρια ευθύνη για μεγάλα τμήματα του προπολογισμού θα μας παρουσιάσουν ε, τον απολογισμό τους. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την συμβολή τους και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά και να συνεργαζόμαστε για την διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Ευχαριστώ, λέει έληξε η συζήτηση για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ξεκινάει η ετήσια διαδικασία χωρίς απαλλαγή Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Σομέτα για την γνωμοδότησή σας. Βεβαίως, ε, χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω επιγόντως κάποια σημεία. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να δώσετε την επαρκή σημασία που σίγουρα θα δώσετε και βασιζόμαστε σε εσά στην έκθεση του συνεδρίου και πιστεύουμε ότι οι συστάσεις οπωσδήποτε θα καταλήξουν σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε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 Ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Okay. Yes, he's there. Yeah, liebe... Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημέρης σας διάταξης. Θα ήθελα να πρότεινα λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω λοιπόν στους συναδέλφους που συνεχίζουν να συζητούν να βγουν από την αίθουσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ λοιπόν όσου συνομιλούν να βγουν από την αίθουσα. Επόμενο θέμα, ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου 6 κάθος 2012 πρόκειται για την ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκο-κυπριακή κοινότητα. Εισηγητής ο κύριος Κάλφιν. τον οποίο παρακαλώ να μας παρουσιάσει το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια έκθεση που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, που συνέταξε το ελεγκτικό συνέδριο και καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Κύπρο. Η ενίσχυση αυτή βασίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2006 και μέχρι στιγμή έχει, ε, υπάρχουν, προβλέπονται γύρω στα 300.000 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορα προγράμματα. Ο στόχος της ε, έκθεσης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής ενίσχυσης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και πιστεύω ότι το ελεκτικό συνέδριο προέβη σε μια πολύ λεπτομερή μελέτη αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει να πούμε ευθύ εξ αρχή ότι η συζήτηση της ενίσχυσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα θέτει όχι μόνο μηγός ε, θέματα που αφορούν τον προπολογισμό και την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Όπως ε, μπορείτε να φανταστείτε, πρόκειται για να θέμα που συνδέεται άρρηκτα με πολύ ευαίσθητα πολιτικά θέματα, αποφάσεις, θέματα που αφορούν ε, ε, την γλώσσα. Και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι και το ελεκτικό συνέδριο στην αξιολόγησή του εκλήθη να αντιμετωπίσει ορισμένα θέματα που δεν άπτονται το δικό του αρμοδιοτήτων που είναι καθαρά δημοσιονομικές. Είναι δύσκολο να γίνει ένας παραλληλισμός με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει μία μοναδικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντισυμβαλόμενο, την ανάγκη του να ε, δοθεί βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε το 2006 ως προσωρινός ε, κανονισμός που είχε στόχο να ε, βοηθήσει την επανένωση στην Κύπρο. Και αυτή είναι μια απόφαση που λήφθη με βάση αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που θα υποβληθεί από το μέλος γίνεται μία αξιολόγηση των προγραμμάτων υπομελέτη και το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι υπάρχουν ορισμένα ελληματικά σημεία αν κάνουμε σύγκριση με άλλα παρεφερή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο πρόγραμμα ιδιάζων σε σχέση με άλλη είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Μερικές φορές είναι δύσκολο να υπάρξει ένας παραλληλισμός και να υιοθετηθούν μέτρα που έχουν υιοθετηθεί αλλού. Το θέμα έχει σχέση και με την διοικητική ε, ικανότητα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από, πριν από λίγο ε, καιρό υπήρχε μία μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία παρακολουθεί από κοντά τον τρόπο εφαρμογής αυτού του προγράμματος και αυτό αποτελεί μέρος της ε, αντιπροσωπείας Επιτροπής στην Κύπρο. Ο προσωρινός αυτός χαρακτήρας το θέμα, τα θέματα που ε, ε εξωθούν ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην χρησιμοποιήσουν τους γνωστούς μηχανισμούς σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της κυπριακής κοινότητας καθιστούν πολύ δύσκολο αυτό το πρόγραμμα στην αξιολόγησή του. Θα ακούσουμε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, εγώ θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονό ότι η περίπτωση αυτή είναι ιδιάζουσα και δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφαρμογής κάποιου άλλου προγράμματος. Από ορισμένε απόψεις θα μπορούσε να γίνει ένας παραλληλισμός με τις ε, ε, ε, την περίπτωση της Παλαιστίνης. Δεν θα έκανα όμως κάποιο παραλυσμό με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σαφείς γι' αυτό. Και τα, οι προβληματικές περιοχές, τα προβλήματα δεν θα μπορούσαν να επιληθούν εφαρμόζοντας μέτρα που έχουν ισχύσει κάπου αλλού. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι και το ελεγκτικό συνέδριο και η Επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και να τους ε, συγχαρώ για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να καταστήσουν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό το πρόγραμμα αυτό από το 2006 και μετά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο παρακαλώ. Όχι. Οπότε να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 12 Νοεμβρίου, τρέχοντος, 12 ώρα το μεσημέρι. Τώρα να δώσω το λόγο στο συνέδριο. Από το συνέδριο ο κύριος Χόρστοκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά εισαγωγικά για αυτή την ειδική έκθεση του συνεδρίου 6 κάθετος 2012 γιατί τη συνοψίζουν τα έγγραφα που έχετε ήδη ενώπιόν σας. Το συνέδριο έκανε μια, έναν έλεγχο αποδοτικότητας για να δούμε εάν η Επιτροπή διαχειριζόταν την οικονομική ενίσχυση στην τουρκυπριακή κοινότητα αποτελεσματικά. Ο έλεγχο αυτός ήθελε να απαντήσει αυτήν την ερώτηση και μόνον αυτήν. Δεν επιχειρήσαμε να αποτιμήσουμε εάν συνολικά το πρόγραμμα συμβάλλει στον στόχο της επανένωσης της Κύπρου, ούτε επιχειρήσαμε να ασχοληθούμε με τα ευρύτερα θέματα που αφορούν το μέλλον της νήσου. Καταλήξαμε σε ορισμένα θετικά συμπεράσματα. Η Επιτροπή τα πήγε καλά για να αναπτύξει το πρόγραμμα, και γενικά για να διαχειριστεί το πρόγραμμα στις δύσκολες ηθίκες ε, στις οποίες χρειαζόταν να εργαστεί. Δαπανήθηκαν οι πόροι με τρόπο που σε αρκετό βαθμό αντικατοπρίζουν τους στόχους και μερικά θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν. Επίσης, ως συνήθως, καταλήξαμε και σε κάποια λιγότερο θετικά πορίσματα. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αφαλάτωσης, απέτυχε. Και έχουμε αμφιβολίες εάν κάποια προγράμματα ούτως ή άλλως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και αν θα συνεχιστούν, εάν και όταν ε, χρειαστεί να διακοπεί η ενωσιακή χρηματοδότηση και κάνει μια σειρά από με βάση τα διάφορα σενάρια για το μέλλον της νήσου. Αυτά όσον αφορά την έκθεση του συνεδρίου. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε, να στραφώ τώρα στην ε, ε, στο αναθεωρημένο σχέδιο έκθεση που έχετε τώρα ενώπιόν σας. Καταρχάς, ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή και τους συνεργάτες του που αξιοποίησαν τόσο καλά την εργασία του συνεδρίου. Η δική μας έκθεση 6 12 σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται σωστά και αντικειμενικά στην έκθεσή σας. Ωστόσο, ελπίζω ότι η Επιτροπή η δική σας θα με συγχωρήσει που θα τονίσω και τρία σημεία όπου νομίζω το σχέδιο έκθεσης πηγαίνει πέρα από την έκθεση του συνεδρίου. Πρώτον, παράγραφος 11 του κειμένου που έχετε μπροστά σας, που λέει ότι έκτιμα ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον προορισμό των ενισχύσεών της να διευκρινιστεί το ερώτημα του πόσος είναι πραγματικά ο τουρκο-κυπριακός πληθυσμός. Και υπάρχει και μια παρόμοια αναφορά στην ιτολογική σκέψη I. Δεν είναι θέμα του ελεκτικού συνεδρίου να σχολιάσει την ε, πολιτική επιχειρηματολογία που είναι πίσω από αυτή την παράγραφο. Αλλά η ειδική έκθεση του συνεδρίου, που είναι, πιστεύω, η βάση του σχεδίου έκθεσής σας, αφορούσε την εφαρμογή του κανονισμού 389 2006. Ο κανονισμός αυτός δεν έκανε καμία διάκριση του τύπου που περιέχεται σε αυτή την παράγραφο όταν αφορά τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό επιπλέον κάποια βοήθεια του προγράμματος δόθηκε σε μεμονωμένα άτομα για παράδειγμα ενίσχυση σε φοιτητές, υποτροφίες τα περισσότερα δόθηκαν για υποδομές ή ε, για το κοινό όφελος όλων των κατοίκων της περιοχής αυτής. Δεύτερο σχόλιο. Παράγραφος 30 του σχεδίου έκθεσης μπροστά σας. Μοιάζει να λέει ότι τα μεγάλα προγράμματα υποδομών θα μπορεί, μπορεί να ε, υποστηριχθούν περισσότερο από άλλα προγράμματα στο μέλλον. Υπάρχουν θέματα απόδοσης προτεραιοτήτων, τα οποία δεν θα αποφασίσει το συνέδριο, βεβαίως. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι τίποτα στην ειδική μας έκθεση 6 κάθετος 2012 δεν λέει ότι τα προγράμματα υποδομών που θα στηρίξει η Ένωση δεν επελέγησαν σωστά, ήταν αδικαιολόγητα ή ότι τα προγράμματα ε, μεγάλης κλίμακος ήταν ανεπιθύμητα με κάποιο τρόπο. Δεν λέει κάτι τέτοιο η δική μας έκθεση. Ακόμη και αυτό το άτυχο πρόγραμμα αφαλάτωσης, από ό,τι ε, αντιλαμβάνεται το συνέδριο, ανταποκρινόταν σε μια σοβαρή πραγματική ανάγκη στην Κύπρο. Αυτό είναι σαφές στην παράγραφο 14 της ειδικής έκθεσης 6 κάθετος 2012. Τρίτο σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Στην παράγραφο 31 εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια πρέπει να υποστηρίξει και όχι να παρεμποδίσει τη διαδικασία επανένωσης της Κύπρου. Κανείς ε, εχέφρον δεν θα, συμφω... δεν θα με κάτι τέτοιο. Αλλά ίσως αυτή η παράγραφος να δίνει την εντύπωση ότι η ειδική έκθεση του συνεδρίου μοιάζει να λέει ότι η βοήθεια όπως δόθηκε τώρα από την Ένωση μπορεί να παρεμποδίζει την επανένωση. Εάν ούτως έχουν τα πράγματα, είναι λανθασμένη η εντύπωση. Όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, το συνέδριο δεν ασχολήθηκε με το εάν και κατά πόσο και σε τι βαθμό αυτές οι βοήθειες βοηθούν την επανένωση της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας ε, για περαιτέρω βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ωστόκ, για την ξεκάθαρη θέση σας ο υποδιευθυντής από την από τη Γενική Διεύθυνση Διεύθυνσης. Φάγκο, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την, το ελεκτικό συνέδριο και τον κύριο Μπόστοκο για την επεξεργασία αυτού του κανονισμού. Νομίζω ότι είναι σαφέ από τι δύο παρεμβάσει, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του σε ό,τι αφορά την Επιτροπή. Δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμία από τι άλλε κατηγορίε τι οποίε καλείται να διαχειριστεί η Επιτροπή. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό και νομικό πλαίσιο. Συνεπώς χαιρετίζω την αναγνώριση αυτών των ε, θεμάτων από το ελεκτικό συνέδριο και θα καλούσα και το Κοινοβούλιο να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση στο ψήφισμα στο οποίο θα πρέπει να τονίσετε τον τρόπο με τον οποίο επιλαμβάνεται των θεμάτων αυτών το ελεκτικό συνέδριο. Τα σημεία αυτά είναι τρία. Καταρχάς το θέμα της διχοτόμησης του νησιού. Το, γενικό, ότι θέλουμε να διευκολύνουμε την επανόνεση του νησιού και τρίτον ότι οι πολίτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι πολίτες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δώσαμε μία απάντηση στα προβληματικά σημεία που ανέφερε το ελεκτικό συνέδριο και σχολιάσαμε μερικά από αυτά. Μπορώ να φερώ τρία. Καταρχάς αναφερθήκαμε στις διαδικασίες, τις κοινωνικές διαδικασίες και συμβάσεων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, αυτών των θεμάτων από τις Βρυξέλλες. Βελτιώσαμε το συντονισμό μεταξύ των γραφείων στη Λευκοσία και του, της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής, η οποία επίσης έχει την έδρα της στη Λευκοσία. Και βεβαίως περιμένουμε να υιοθετηθεί μια απόφαση ό,τι αφορά το μήκο των συμβάσεων για το προσωρινό προσωπικό, κάτι που συνδέεται με τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή ε, στα πλαίσια του νέου πλαισίου. Μια ένα εκτενέστερο χρονικό διάστημα θα μας επιτρέψει να απασχολήσουμε το προσωπικό και να είναι περισσότερο αποτελεσματικό στη δουλειά του στη Λευκοσία. Θα ήθελα να αφαιρθώ σύντομα σε δύο συγκεκριμένα θέματα, κύριε Πρόεδρε, συντομία. Καταρχάς, το πρόγραμμα για το εργοστάσιο αφαλάτωση της Αλασίου Ήδατος δεν είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που χρηματοδοτήσαμε και απέτυχε. Και απέτυχε για λόγους που εξηγούνται εκτενώς στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Κανένα πρόβλημα για μας είναι πως αυτό. Το βεβαίως το μέγεθος του έργου αυτού ήταν πάρα πολύ μεγάλο, 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δαπανώνται στο νησί. Ήταν ιδιαίτερα λυπηρό το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό που θα μπορούσα να πω σε ό,τι αφορά τα διδάγματα που έχουμε μάθει είναι ότι εξετάζουμε τις δυνατότητες να βρεθεί εναλλακτική, ένας εναλλακτικός τρόπος βοήθειας σε ό,τι αφορά την παροχή ύδατο, που είναι ένα πρόβλημα για το νησί. Δεν είναι εύκολο όμω να διασωθεί αυτό το έργο. Δεύτερον, το θέμα που αφορά την βιωσιμότητα των παρεμβάσεών μα, Ένα θέμα που έθιξε πριν από λίγο ο κύριος Μπόσταξ, στο σημείο 60 της έκθεσης. Αυτό είναι ένα πραγματικό θέμα που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας σε επικοινωνία με τους ομολόγους μας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν στα πλαίσια του νομικού και διοικητικού πλαισίου για να μπορέσουμε εμείς με τη σειρά μας να συνεχίσουμε ε, τη συνεργασία μας σε αυτό το έργο. Το λεκτικό συνέδριο με κατά τον ίδιο τρόπο αναφέρεται, τονίζει στο θέμα της έλλειψης προβλεψιμότητας της ενίσχυσης. Όπως τα αξιότιμα μέλη γνωρίζουν, ο κανονισμός ο ίδιος του 2006 δεν ε, θα εκπνεύσει τη στιγμή που θα υπάρξει μια ρύθμιση. Ελπίζω να γίνει σύντομα αυτά, αλλά δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Τα χρήματα που έχουν δοθεί από την αρχή του προπολογισμού έχουν τελειώσει. Και συνεπώ η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθεί κάθε χρόνο να προσπάθει τα χρήματα από την αρχή του προπολογισμού, τα οποία θα πρέπει να αποσύρονται από το απόθεμα. Και αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο για μα την Επιτροπή να καταφέρει έναν εκ των προτέρων σχεδιασμό κάθε χρόνο εξαρτώμεθα από την καλή θέληση των αρχών του προϋπολογισμού. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και υποβάλαμε μια πρόταση για να ρυθμιστεί το πλαίσιο, στο θέμα αυτό στα πλαίσια του πολιετούς ε, πλαισίου και θα είναι πολύ πιο εύκολο για μας να διαχειριστούμε τα προγράμματα σε μια πιο μακρόπνοη βάση. Επουδενή δεν θέλω να δημιουργήσω την εντύπωση ότι θέλουμε να συνεχιστεί περισσότερο το πρόγραμμα. Το αντίθετο, όσο πιο νωρί τελειώσει, τόσο το καλύτερο, γιατί σημαίνει ότι έχουν διευθετηθεί τα πράγματα στο νησί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεση, ε, μπορώ ε, να είμαι πολύ σύντομο. Συμφωνώ με όλα τα σημεία που ανέφερε ο κύριος Μπόστοκ. Ε, θα ήμουν ε, ιδιαίτερα ευτυχής αν το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να περιοριστεί σε θέματα που αφορούν τον ίδιο τον κανονισμό και αν θα μπορούσε να αποφύγει, να ε, προσθέσει και άλλα στοιχεία που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του συγκεκριμένου κανονισμού. Το θέμα των επίκων στο νησί είναι ένα θέμα ε, καθοριστική σημασία και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τι διαπραγματεύσει. Αυτό όμω είναι ένα θέμα που εμεί δεν μπορούμε να λύσουμε στα πλαίσια της, του συγκεκριμένου αυτού κανονισμού ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει για την παράγραφο 30 και 31. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξή Μου είπαν ότι η επόμενη έκθεση ήταν να τη συζητήσουμε μετά, να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη, δηλαδή αν δεν έχετε αντίρρηση. Πάντως προς το παρόν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτής της ειδική έκθεσης. Δεν θέλει όμως κανείς το λόγο γι' αυτό για να συνοψίσει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπόστοκ και τον ε, αναπληρωματικό γενικό διευθυντή του. δεν διαφέρουμε στην προσέγγιση μας. Πρέπει να τονίσουμε δύο πολύ σημαντικές αρχές. Πρώτον, στην ορολογία και στις, στη διατύπωση. Είχε ήδη συμφωνηθεί μια διατύπωση που να χρησιμοποιείται και από το Συμβούλιο και από τα ψηφίσματά μας. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο θέμα που περιγράφει αυτή η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και όχι και άλλα διαπλεκόμενα. Αυτό θα υποστηρίξω εγώ και στην τελική μορφή της έκθεσής μου. Για τα σχόλια του κυρίου Μποστόκ τώρα ως προς το μέγεθος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση από αυτήν των ενωσιακών κονδυλίων ίσως να έχει κάποια σημασία το μέγεθος της κοινότητας αλλά δεν είναι κάτι απόλυτο. Θα ληφθεί υπόψη τέλος πάντων. Όσο για τα προγράμματα μεγαλύτερης εμβέλειας, μεγαλύτερης κλίμακας, δυστυχώς το σπουδαιότερο από αυτά απέτυχε και αυτό όχι γιατί δεν έκανε αρκετές προσπάθειες η Κομισιόν ή για οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους έλλειψη, αλλά λόγω πολιτικών δυσκολιών. Η Κομισιόν παρόλα αυτά μπόρεσε να το διορθώσει αλλά μετά ο συμβαλόμενος αρνήθηκε. Η Κομισιόν πάντως έκανε ό,τι μπορούσε. Αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα του τι συμβαίνει και στην ίδια την έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου αναφέρεται το θέμα της ιδιοκτησίας γης μεγάλο τμήμα της οποίας 78% ανήκει σε Ελληνοκύπριους. Πρέπει όμως οι συνομιλητές μας να είναι αρχές τις οποίες να αναγνωρίζουμε και αφού μιλάμε νομικά βλέπουμε τα πράγματα ως ένα κυπριακό κράτος με ορισμένες περιφέρειες που δεν ελέγχει η κυβέρνηση. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει ομαλά δεν μπορεί να είναι όλα ομαλά σε όλα μας τα προγράμματα αφού είναι έτσι τα πράγματα. Και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν ισχύει. Γι' αυτό θεωρώ ότι το πρόγραμμα ήταν πολύ αποτελεσματικό προς την κοινωνία των πολιτών, την ελεύθερη διακίνηση, τους αγνοούμενους, θέματα ιστορικών τοποθεσιών κλπ. Όλα αυτά τα προγράμματα ήταν πολύ επιτυχή και αποτείω εδώ φόρο τιμής στην Κομισιόν για την επιτυχία αυτή. Αλλά λόγω των θεμάτων που σχετίζονται με το Κυπριακό θα έχουμε δυσκολίες με οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας και στο μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα η ευρωπαϊκή βοήθεια να επικεντρωθεί στους τομείς όπου αποδείχτηκε ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα. Συμφωνώ βέβαια με τον κύριο Μποστόκ. Δεν νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο εμποδίζει την επανένωση και άλλα τέτοια που ακούστηκαν. Νομίζω ότι γενικά το ελεγκτικό συνέδριο βοηθάει, υποβοηθάει την ενοποίηση της Κύπρου, την επανένωση. Τέλος, μία σύσταση της έκθεσής τους είναι και αυτή που μας είπε η ίδια η Κομισιόν. Προς στιγμή, μα μέχρι τώρα υπάρχει ένας μηχανισμός που είναι βράχη πρόθεσμης διάρκειας για τους τροκοκύπριους. Ενώ το ελεκτικό συνέδριο έχει εξετάσει και τις πιθανότητες επανένωσης της Κύπρου αλλά αυτό δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτά, να πάρουμε υπόψη μας υποθέσεις και σενάρια. Ελπίζουμε μεν να λυθεί το πρόβλημα σύντομα, αν και τόσα χρόνια χρονίζει. Και δεν θα λάβουμε υπόψη μας τα σενάρια της επανένωσης. Θα βασιστούμε στην υπόθεση ότι μπορεί να γίνει η επανένωση, αλλά το πρόγραμμα θα παραμείνει ουδέτερο και θα υποβοηθήσει την επανένωση αν συμβεί αντί να υποθέτει ότι θα γίνει να, σαν προϋπόθεση δηλαδή. Πιο μακροπρόθεσμα λοιπόν προγράμματα και μεγαλύτερης κλίμακας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Απ' την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι de facto παίρνουμε σαν βάση τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου. Όπως και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και στη δική μου, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον κανονισμό AID, AID που διέπει αυτή τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Δεν θα προδικάσουμε όμως τίποτα δεν θα προκαθορίσουμε αν ένα πρόγραμμα θα είναι βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο κτλ. με βάση την επανένωση ή μη της Κύπρου. Αυτό πρέπει να προσέξουμε στη διατύπωση και να βασιστούμε σε αυτές τις δύο αρχές, τις διατυπώσεις που έχουν συμφωνηθεί και όσο το δυνατόν να περιορίσουμε και τους στόχους μας σε αυτά που λέει η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Κάλφιν. Διαμαρτυρήθηκε συνάδελφος ότι τον παρέβλεψα. Αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει συχνά εδώ. Αλλά παρακαλώ. Παρακαλώ. Ρωτάω λοιπόν όλους του συναδέλφου που θέλουν να μιλήσουν για την Κύπρο να μου πούν εάν το θέλουν. Κάποιον παρέβλεψα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άλλο. Ο κύριο Ζώνικ, παρακαλώ λοιπόν. Ε, έχει το λόγο και μετά χρειαστεί πάλι ο κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ προσοχή την παρουσίαση αυτή της έκθεσης του Ελληνικού Συνεδρίου όπως επίσης και την, ε, τις άλλες παρουσιάσεις. Καταλήγω λοιπόν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνέχιση της χρηματοδότησης πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη η δέσμευσή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό πρέπει να εγγυηθούμε στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν θέλω να πω ότι αυτή η εγκατάσταση αφαλάτωση είναι ιδιαίτερα λυπηρό το ότι απέτυχε. Ιδιαίτερα λυπηρό το πρόγραμμα αυτό ε, είχε εγκριθεί στο σωστό πολιτικό επίπεδο. Το είχαμε συζητήσει ή θα έπρεπε να το συζητήσουμε και στα πλαίσια των συζητήσεών μας ε, ένταξη με την Τουρκία. Θα έπρεπε να συζητηθεί, λυπάμαι που για λόγους πολιτικού ε, μπλοκαρίσματος δεν μπόρεσε να προωθηθεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Ζόνικ. Θέλετε να πείτε κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Λέει ο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντής για τη Διεύρυνση. Υπάρχει ένα θέμα με τον τουρκικό στρατό για αυτήν την εγκατάσταση αφαλάτωσης στην πρώτη φάση του προγράμματος. Αυτό καθυστέρησε τα θέματα. Στο τέλος επελήθη αυτό το θέμα. Δηλαδή ο στρατός επέτρεψε να συνεχιστούν οι εργασίες. Αλλά σε αυτή τη φάση και μετά από τόσε καθυστερήσει, η τεχνική εταιρεία που την είχε αναλάβει, ο ανάδοχο που ήταν από την ε, Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε ότι δεν τον ενδιαφέρει πια αυτό το έργο. Οπότε αυτό τελικά ήταν ε, η τελική εγκατάλειψη αυτού του προγράμματος, η τελική αποτυχία του. Το θέμα λοιπόν με τον τουρκικό στρατό ε, επελήθη. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρφιν δεν θέλει το λόγο, οπότε κλείνουμε την συζήτηση για το θέμα αυτό σε αυτή τη φάση. Υπάρχει δυνατότητα, όπως είπα, υποβολής τροπολογιών 12 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Η έκθεση θα ψηφιστεί στις 26 Δεκεμβρίου με βάση τον ε, τρέχοντα προγραμματισμό εργασιών μας. Επόμενο θέμα λοιπόν, συμφωνείτε την έκθεση του κυρίου Στάς να την ε, συζητήσουμε πριν από το επόμενο θέμα, όπως ζήτησε ο κ. Στάς. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον εδώ ο εισηγητής. Είναι η ειδική έκθεση 13-2012 και ιδιαίτερα για το θέμα της διαδικασίας για τα τελωνία σε σχέση με το ΦΠΑ. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Στάς και από πλευρά ελεκτικού συνεδρίου είναι εδώ ο διευθυντή Μάρτιν Τσβίκλ, που είναι ο αρμόδιο. Οπότε, να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο. Κύριε Τσβίκλ. Μπορείτε παρακαλώ από πλευρά σας να μας παρουσιάσετε τα βασικά θέματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω σύντομα τα κυριότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έκθεσής μας. Επίσης στην παρουσίασή μου θα παρουσιάσω λιγάκι τι έγινε από τότε που γράφτηκε η έκθεση γιατί υπήρξαν ορισμένε εξελίξεις και είμαι σίγουρος ότι αργότερα θα συζητήσουμε και με τον εισηγητή. Πρέπει να γνωρίζουμε βεβαίως ότι το ΣΠΙΛ είναι πρόγραμμα που το CP42. Αφορά κυρίως προβλήματα μεταφοράς ΦΠΑ. Οι εισαγωγές μπορούν να παραμένουν σε μια χώρα μέλος αν δεν έχει πληρωθεί ΦΠΑ και ίσως να επιτρέπεται και η κατανάλωση τους χωρίς καταβολή ΦΠΑ εκτός αν δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες βέβαια. Ο κύριος στόχος του ελέγχου ήταν να δούμε αν η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη εφήρμοσαν ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για να αποφευχθεί η διαφυγή. Και για να γίνει αυτός ο έλεγχος καταρτήσαμε ένα πρότυπο με βάση προηγούμενα προγράμματα για την ε, αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ και επισκεφθήκαμε 7 χώρες μέλη, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία διότι οι χώρες αυτές αντιπροσώπευαν το 68% της αξίας των εισαγωγών με βάση αυτή τη διαδικασία κατά το έτος που αναφοράς. Για κάθε χώρα μέλος διαλέξαμε 20 με 30 εισαγωγές Ο στόχος του δειγματοληπτικού αυτού ελέγχου ήταν να δούμε πώς εφαρμόζεται το πρότυπο του ΕΚΑ μετά αν χρειάζεται καμία συμπλήρωση και τρίτον Εάν υπολογίστηκε και αναφέρθηκε η πληρωμή μη του ΦΠΑ των εισαγωμένων στα εισαγόμενα αγαθά. Διαπιστώσαμε δε τα εξής. Πρώτον, για τις χώρες μέλη διαπιστώσαμε ότι δεν διασφαλίζουν πάντοτε τις συνθήκες εξαίρεσης από τον ΦΠΑ. Δεύτερον, δεν γνωστοποιούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές εάν πληρώθηκε όχι ο ΦΠΑ και τρίτον, δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που έχουν για να ταυτίσουν και να καταπολεμήσουν την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. Θελήσαμε να καταλήξουμε σε αριθμού συγκεκριμένους και το συνολικό ποσό της απώλειας ΦΠΑ ήταν 2,2 δισεκατομμύρια για το 9. Θέλησαμε να αναλύσουμε τι ακριβώς σημαίνει το ποσό αυτό και καταλήξαμε ότι αντιπροσωπεύει το 29% του συνολικού ΦΠΑ. Σε επίπεδο κομισιών διαπιστώσαμε ότι αν και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών με τα διάφορα νομοθετικά πρότυπα που έχει προβλέψει και ιδιαίτερα την οδηγία ΦΠΑ πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες γιατί κατ' εμάς το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν διασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή των εξαιρέσεων αυτών από το ΦΠΑ. Δηλαδή οι τελωνιακές αρχές δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε. Ή εναλλακτικά δεν δίνονται οι πληροφο σχετικές πληροφορίες στις φορολογικές αρχές των χωρών μελών. Και τα δύο αυτά τα εκμεταλλεύονται οι απατεώνες Στη βάση του ελέγχου μας κάναμε 8 συστάσεις πολύ λεπτομερείς, αλλά κυρίως 3. Θα έπρεπε νομίζω με Κομισιόν πρώτον να προτείνει την τροποποίηση της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη να χορηγούν και να ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά μία συναλλαγή. Οι χώρες που εισάγουν τα προϊόντα αυτά πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά και δεύτερον λέει ο Μίλητης να υπάρξει σε ενωσιακό επίπεδο ένα ενιαίο πρότυπο ελέγχων που να μας επιτρέπει να κάνουμε αυτόματη και πλήρη ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών. Το λεγόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Και τρίτον και τελευταίον, να ενθαρρύνει το Συμβούλιο να τροποποιήσει την οδηγία του ΦΠΑ ώστε ο εισαγωγεύς να είναι υπεύθυνο για, ε, για τον ΦΠΑ. Μάθαμε με χαρά ότι και ο κύριος στάσος ηγητής της σχετικής έκθεσης, δέχεται όλες μας τις συστάσεις. και ότι η τροποποίηση για την οδηγία του ΦΠΑ γίνεται και αυτή δεκτή. Επίσης, γραπτός σας είχαμε πληροφορήσει για ορισμένες επιπτώσεις που είχε η έκθεση αυτή η Πορτογαλία, η Σλοβενία ζήτησαν παρόμοιο έλεγχο να εφαρμοστεί και σε χώρες εκείνες τον Μάρτιο φέτος εξεδόθη μία γνωμοδότηση που λάμβανε υπόψη της αυτήν την ειδική έκθεση και ζήτησε από την Κομισιόν να τροποποιήσει περαιτέρω το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και το ΕΚΟΦΗΝ επίσης με τη σειρά του είπε ότι μέτρα βελτίωσης του ρυθμιστικού αυτού πλαισίου, του νομοθετικού αυτού πλαισίου έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται μεν, αλλά ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται για αυτό το θέμα και να προσέχουν περισσότερο το θέμα της ε, φοροαποφυγής σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία CP42. Και το Eurofisc το εξετάζει το θέμα, άρα έχουν υπάρξει ενδιαφέρουσες εξελίσεις και μεγάλο ενδιαφέρον και θα μπορούσε κανείς να καταλήξει ότι ναι μεν η απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος εάν η διαδικασία CP42 μπορεί να ταυτίσει τις ε, αποφυγές ΦΠΑ η απάντηση είναι όχι αλλά οι συστάσεις που κάνουμε θα μπορούσαν να καταλήξουν σε θετική απάντηση, σε καλύτερη δηλαδή πρόληψη της ΦΠΑ αποφυγής. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσβίκλη για την εισαγωγή σας. Θα θέλει το λόγο εισηγητής τώρα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο ανταλλάξαμε τις ε, απόψεις μας. Ήταν θαυμάσια αυτή η έκθεση αυτή, πολύ συγκεκριμένη, με πρακτικά απορίσματα. Τονίστηκαν τα σημεία που προκαλούν τριβές εδώ. Γίνονται 7 συγκεκριμένες ε, συστάσεις. Θαυμάσια εργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε όμως συνολικά το πλαίσιο, να το σκιαγραφίσω. Ξέρουμε ότι είμαστε σε δύσκολες ε, Ε, συνθήκες και ότι χρειάζεται σε πολλά σημεία να σφίξουμε το ζωνάρι. Ξέρουμε ότι ε, η φορολογική απάτη υπολογίζεται σε 200-250 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποφυγή και η απάτη του ΦΠΑ ε, υπολογίζεται σε περίπου 100 δις. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρή υπόθεση, ιδιαίτερα σοβαρή. Βεβαίως εξετάσαμε προσεκτικά τον κανονισμό και θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία το 2009 είχε ως αποτέλεσμα 2,2 δις με βάση αυτόν τον έλεγχο σε 7 χώρες. Άρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν το θέμα αυτό και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η έκθεση. Σε κάποιο σημείο της ε, έκθεσής μου τονίζω ότι υπήρξε μία μελέτη που ε, χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι, ότι η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα που θα έπρεπε να είχαμε από αυτόν τον πόρο ε, και τα πραγματικά έσοδα ε, είναι της τάξης του 12% και στις νότιες χώρες μέλη που έχουν τα σοβαρά προβλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερη. 30% στην Ελλάδα, 22% στην Ιταλία. Γι' αυτό καλωσορίζω αυτή την έκθεση. Την καλωσορίζω ιδιαίτερος. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου καταδεικνύει σαφώς ότι φταίει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες βελτιώσεις. Και παράλληλα τονίζει το ελεγκτικό συνέδριο ότι μέσω των ε, τελειωναϊκών ελέγχων πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. δεν γίνεται σωστά ο έλεγχος, δεν απαιτείται η σωστή τεκμηρίωση. Η ε, προσπάθεια συλλογής του ΦΠΑ δεν έχει αλλάξει εδώ και αρκετά χρόνια. Πρέπει να αλλάξει. Υπήρξε μια πράσινη βίβλος, έχουν γίνει μια σειρά μελέτες και αυτό το αναφέρω σε κάποιο άλλο σημείο της εκθεσής μου. Συζήτησα ε, κατά πολύ και επανειλημμένα με προσώπους τελωνιακών και φορολογικών αρχών που με έπεισαν μου είπαν ότι ήδη έχουν γίνει πολλά και σε αυτούς θα ήθελα να δώσω το λόγο. Παρακαλώ, πείτε μας τι έχετε κάνει συγκεκριμένα και τι πρέπει ακόμη να επιτελεστεί, ούτως ώστε και εμείς να ασκήσουμε πίεση, να διατηρήσουμε την άσκηση πίεσης. Θα έπρεπε λοιπόν και το προτείνω μέσα στο 2013 να υπάρξει ένα follow-up, να εξακολουθήσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, ούτω ώστε να μελετήσουμε προσεκτικά το θέμα αυτό. Αυτά λοιπόν που μα υπέβαλε το Ελληνικό Συνέδριο, τι συστάσει και δράσει που προτείνει, να συνεχίσουμε να πιέζουμε για την εφαρμογή του, ούτω ώστε επιτέλου να εφαρμοστούν. Από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν επίσης θα ήθελα να ακούσω τι δυνατότητες υπάρχουν μέσω της καλύτερης χρήσης του ε, Eurofisk. Βεβαίως, συνεργάζονται κάποιες χώρες μέλη μαζί του, αλλά δεν συμμετέχουν όλοι, αυτό το γνωρίζω σαφώς. Μήπως θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να συνδέσουμε όλα τα κράτη-μέλη στις εργασίες αυτού του σώματος, ούτως ώστε το θέμα αυτό να προωθηθεί περαιτέρω. Σε σχέση πάντα με την ε, τελωνιακή διαδικασία 42. Είπα λοιπόν ήδη ότι υπάρχουν 7 συστάσεις που μας υπέβαλε το Λεκτικό Συνέδριο, τις υποστηρίζω εκπεφρασμένα και επιπλέον, επιπλέον, σε ένα σημείο της εκθεσή μου, θεωρώ ότι είναι υπεύθυνοι και οι ε, έμποροι. Εάν δεν δηλώσουν σωστά στο τελωνίο ή εάν δεν κάνουν καθόλου δήλωση στο Τελωνείο πρέπει και αυτοί να θεωρηθούν υπεύθυνοι. Πρέπει να τονιστεί αυτό, είναι σημαντική πρόταση και καλό την Κομισιόν να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αυτή την ε, πρότασή μου. Καλό την Κομισιόν να κάνει περαιτέρω συγκεκριμένε προτάσει. σω θα ήταν σκόπιμο, κύριε Πρόεδρε, να, κάνουμε, να δώσουμε το λόγο και στην Επιτροπή για να μα πει πώ αντιδρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγητά. Αυτό θα κάνουμε. Αλλά παρακαλώ και τους άλλους συναδέλφους που έχουν ερωτήσει προς την Κομισιόν να τις θέσουν τώρα. Σάλφος Γκάια. Α, θέλει να κάνει σχόλια. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Όχι. Οπότε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο οποίος είναι ο Μύρος Λαβζιλίνσκι από την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι προσεκτικά εξετάσαμε την έκθεση, δεχτήκαμε τις συστάσεις και ήδη ένα μεγάλο μέρος της εργασίας έχει γίνει. Βεβαίως δεν είναι πολύ ευχάριστο το να ακούει κανείς ότι κάτι θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ καιρό πριν. Παρόλα αυτά θέλω να πω ότι η δουλειά έγινε, δεν είναι πάντοτε πολύ γοργή η ρυθμή και σε επίπεδο νομοθετικό αλλά και σε επίπεδο εφαρμοστικό. Έχω έρθει με διάφορους συναδέλφους. Εγώ θα επικυρώσω την προσοχή μου στο θέμα των τελωνίων και μετά με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε θα ζητήσω από τον συνάδελφό μου να μιλήσει ε, για το θέμα του ΦΠΑ. Ο συνάδελφός μου είναι τμήματάρχης. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία στα τελωνία και αυτό που καταλάβαμε από τις συστάσεις και το είχαμε καταλάβει εξάλλου και στο παρελθόν ότι το βασικό πρόβλημα από την άποψη των τελωνίων αφορούσε την επικοινωνία μεταξύ των τελωνιακών και των φορολογικών αρχών. Και Αφού γίνουν τα πάντα, τίθεται το θέμα του ελέγχου των διαδικασιών. Πώς όλα αυτά εφαρμόζονται πρακτικά στις χώρες μέλη. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι από πλευρά τελωνίων η Επιτροπή και οι χώρες μέλη περάτωσαν το Δεκέμβριο του 2009 μία ρύθμιση διοικητική σε ό,τι αφορά την σωμάτωση του αριθμού του ΦΠΑ στις τελωνιακές διασαφήσεις. Αυτή η συμφωνία, αυτό το κείμενο αναφέρει ότι το ΦΠΑ των ατόμων που αναφέρονται στη διαδικασία 42 θα πρέπει να εντάσσονται στο σημείο 44 των διασαφήσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένου κώδικες. Δηλαδή, το είδος της, ε, του προορισμού και το είδος των αγαθών έχει ήδη κωδικοποιηθεί στο τετραγωνίδιο 44. Αυτό, αυτή η ρύθμιση συμπεριλήφθη στις τροπολογίες που υπευλήθησαν στον κανονισμό της Επιτροπής 756 του 2012. Αυτό που κάναμε, αφού προβήκαμε στην ανάλυση της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου, είναι ότι τονίσαμε για μία ακόμα φορά όσα περιέχονται στην νομοθεσία, αλλά ενδεχομένως δεν ήταν απόλυτα σαφές. Δηλαδή, ακόμα και διατρέχοντας τον κίνδυνο να επαναλάβουμε τις ίδιες νομικές διατάξεις, θελήσαμε να καταστήσουμε απόλυτα σαφές αυτό και να αποφύγουμε περιπτώσεις όπου ένας συγκεκριμένος εμπλεκόμενος στη συγκεκριμένη διαδικασία μας πει ότι κάτι δεν είναι σαφές. Συνεπώς, οι ευθύνε των τελωνιακών αργών είναι πλέον σαφείς. Από την άποψη της εφαρμογής προσπαθούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ των τελωνιακών αξιωματούχων και των αξιωματούχων των ε, φορολογικών υπηρεσιών στις χώρες μέλη. Δεν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα, δεν μπορούμε να ε, κάνουμε ένα κοινό σύστημα τελωνίων και ΦΠΑ. Συνεπώς, παραμένουμε στα πλαίσια της ανακοίνωσης που στείλαμε στις χώρες μέλη και βασιζόμαστε στους συναδέλφους που ασχολούνται με το ΦΠΑ να φροντίσουν έτσι ώστε η, ανακοι... η... η επικοινωνία μεταξύ της χώρας μέλους όπου ε, ε, ε, έφτασαν τα αγαθά και της άλλης χώρας μέλου όπου θα έπρεπε να καταναλωθούν τα αγαθά θα είναι μια επικοινωνία αποτελεσματική. Ύστερα αρκετές πρωτοβουλίε ελήφθησαν από πλευράς ΦΠΑ. Με την άδειά σα, λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα επιθυμούσα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου τον Τόμ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά γενικά λόγια. Ήμουν υπεύθυνο στον τομέα αυτό, στον τομέα μέσων κατά την καταπολέμηση της απάτης και γενικά θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα θέματα απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και αυτό που μας απασχολεί είναι γενικά η απάτη σε θέματα ΦΠΑ. Και πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια ανακοίνωση για διάφορε δράσει που θα επιθυμούσαμε να ληφθούν για να απανταχθεί το θέμα τη ε, ε, φορολογική απάτη. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα. Το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το θέμα και όπου είναι αναγκαίο υποβάλλουμε τις αναγκαίες προτάσεις, νομοθετικές προτάσεις για τις χώρες μέλη για να μπορέσουν να δράσουν. Θα ήθελα να τονίσω τη διάκριση, τη σαφή διάκριση που υπάρχει το ρόλο και την ευθύνη τη Επιτροπή από τη μία πλευρά και το χωρό μελών από την άλλη. Εμεί δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή, για την ίσπραξη του ΦΠΑ. Οι χώρε μέλη είναι υπεύθυνε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό βάσει των οποίων οι διάφορε αρχέ συνεργάζονται μεταξύ του έτσι ώστε να γίνεται σωστά η δουλειά. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ποιο είναι υπεύθυνο και δεν είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα τη διαδικασία ε, ξέραμε ότι υπήρχε μία έλλειψη στον τομέα αυτό, στη διαδικασία αυτή και αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα για να αφαιρθώ στα όσα ε, αναφέρθηκαν στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, ε, τροπολογήσαμε την νομοθεσία έτσι ώστε τα αγαθά που εισάγονται με βάση τη διαδικασία 22 εντάσσονται στο σωστό σύστημα ανταλλαγής ΦΠΑ. Δεύτερον, δημιουργήσαμε το δίκτυο Eurofist, με το οποίο αναφέρθηκε ο εισηγητής. Αυτό είναι ένα δίκτυο αξιωματούχων στις χώρες μέλη που ασχολούνται με συγκεκριμένες πληροφορίες δυνητικών περιοχών όπου έχει διαπραχθεί απάτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα συγκεκριμένο τομέα που αναφέρεται με τη διαδικασία των τελωνίων 22. Customs 22. Ε, ε, ε, η Επιτροπή δεν είναι μέλος της Eurofish. Όπως είπε, πρόκειται για μια διακυβερνητική κατάσταση όπου εμείς δίνουμε στην ουσία μια στήριξη. Και εξετάζουμε τον τρόπο λειτουργίας και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα συστήματα που επιτρέπουν σε αυτό το δίκτυο να λειτουργήσει όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματικά. Και πάλι όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι χώρες μέλη έχουν ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο το έθεσαν αυτό το δίκτυο αποκλείοντας την Επιτροπή. Γιατί πάντοτε μας θυμίζουν ότι είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας δεν ξεχνάμε ποτέ να μας το πούν. Ένα από αυτά που θα κάνει το Eurofist σε πλαίσια της διαδικασίας Customs του αιτητού είναι το θέμα του περιγράμματος που είπαμε πριν από λίγο και αυτό είναι κάτι που παρακολουθούμε από κοντά και προσπαθούμε να ε, ε, εξετάσουμε. Άλλα θέματα που θα μας ικανοποιούσε η στήριξη του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εθελοντική φάση ε, της συμμετοχής των χωρών μελών σε αυτόν τον τομέα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι, είναι καταβούληση, είναι θελοντική η συμμετοχή, δεν είναι υποχρεωτική σε αυτό το τομέα. Βεβαίω και αυτό θα θέλαμε να το υποστηρίξουμε. Το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρθηκε στο θέμα της υπάρχουσας ε, πρότασης που αφορά τη συνυπευθυνότητα. Αυτό έχει τεθεί στο Συμβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η ε, υποστήριξή σας και πραγματικά θα απευθύναμε έκκληση στους αρμόδιους να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, δεν είπαμε ότι θα αναφερθούμε όσο γίνεται πιο συχνά σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, πιστεύω ότι μερικές από τις συστάσεις που έγινα στο σχέδιο έκθεσης είναι κάπως ουτοπικές από την άποψη της Επιτροπής. Δεν έχουμε τους πόρους και την ικανότητα να αναφερόμαστε δύο φορές το χρόνο. Εμείς θα υποβάλουμε μια έκθεση του άρθρου 12 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται η ίσπραξη των ίδιων πόρων. Έχουμε αποφασίσει να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο, το στείλαμε στις χώρες μέλη και εκεί ζητάμε να μας πούν τι μέτρα ακριβώς υιοθέτησαν για να εφαρμόσουν διαδικασία Customs 22 τι ε, μέτρα λαμβάνουν έτσι ώστε να μπορούν οι ε, τελωνιακές αρχές ε, να έχουν πρόσβαση στην βάση του ΦΠΑ και να ελέγχουν την ακρίβεια. Ελπίζω ότι με την έκθεση που θα υποβληθεί του χρόνου θα μπορέσουμε λεπτομερώς να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα των ευρημάτων μας καθώς και για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστάσεων και τη διαδικασία Customs 22. Ευχαριστώ. Yeah, thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Ένα άλλο ηγεστής το λόγο. Γκάια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τονίζω πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η ειδική έκθεση και με βάση και την πολιτική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε πρέπει οπωσδήποτε να εξαγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα. Στη συζήτηση προηγουμένως για την απαλλαγή δεν το τόνισα αρκετά συγκεκριμένα, αλλά εγώ θα επιθυμούσα ιδιαίτερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, όπου είμαστε σε ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου από τη μία και κρατών, και κρατών μελών από την άλλη, θα με ενδιέφερε λοιπόν να διαπιστώσουμε και όπου το αντικείμενο της συζήτηση είναι πόσα θα μας δοθούν, είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι έσοδα που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα έσοδα από το ΦΠΑ, σε τι βαθμό πραγματικά εισπράττονται και αξιοποιούνται. Έχει λοιπόν πολιτική σημασία να τονίσουμε σαφώς πώς έχει κατάσταση για να ασκήσουμε επίσης τα κράτη-μέλη. Εφόσον πρόκειται για συλλογή ιδίων πόρων και για τους ίδιους και για την Ένωση να μην επιτρέπουμε τέτοιες ε, προχειρότητες. Με εντυπωσιάζουν αυτά τα ποσοστά που αναφέρθηκαν. 2,2 δις δεν πρόκειται για πενταροδεκάρες. Με τέτοια ποσά μπορεί να κάνει κανείς πολλά. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους θερμότατα να δουν πως σε συνδυασμό με την Κομισιόν θα μπορούσαμε με βάση αυτά που μάθαμε από το Ελληνικό Συνέδριο να τονίσουμε τι προβλήματα υπάρχουν στα έσοδα. Να δούμε λοιπόν εάν οι υπάρχουσες διαδικασίες για τη συλλογή εσόδων της Ένωσης δεν θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Με βάση αυτή την έκθεση που μόλις άκουσα και με βάση ε, την έκθεση που έκανε συνολικά για το θέμα των τελωνίων Μπάρτ πριν από μερικού μήνε, είναι πιστεύω ένα θέμα που θα μπορούσε να μα απασχολήσει. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Το λόγο λέει ο πρόεδρο για το θέμα αυτό. Όχι. Α, παρακαλώ. Α, α βλέπω ότι συμφωνείτε. Κυρία Γκρέσλε, δεν θέλετε το λόγο. Ωραία. Οπότε ο εισηγητή. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα σημειώνω την αντίδραση της Κομισιόν προς την ρεαλιστική ερώτηση που είχα θέσει. Επίσης, βλέπω ότι η έκθεση για το άρθρο 12 θα γίνει φέτος και ο κανονισμός για το 42 και παρακαλώ να μας, τα δώσετε, να μας τις δώσετε αυτές τις εκθέσεις στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Για μας θα ήταν πολύ χρήσιμα και συγκεκριμένα για την έκθεσή μου, διότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε την πίεση και την πληροφόρηση για το τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Μα μόνο να συμφωνήσω μπορώ, λέει ο Πρόεδρος, με αυτά που είπε ο εισηγητής. Δεν θα πρέπει να χάσουμε από την προσοχή μας το θέμα αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Κομισιόν. Τροπολογίες μέχρι 12, 11, 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε λοιπόν την ημέρησια διάταξη, οπότε κάτι ακόμη να σας πω. Για ένα θέμα που έχουμε πριν την ημέρησια διάταξη, της κατεξιοδότηση πράξης. επί του οποίου να σας πω το εξής. Στις 29 Οκτωβρίου 2012 το Κοινοβούλιο έκανε τις μεταφράσεις για τον κανονισμό για τους κανόνες εφαρμογής του Γενικού Προπολισμού της Ένωσης. Όλο αυτό το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτές οι κατεξουσιοδότηση πράξεις περιέχουν μια σειρά κανόνων για τη χρήση των δημοσιονομικών κανόνων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Για παράδειγμα, ο κανονισμό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρατόμ 966 κάθε 2012 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 Οκτωβρίου 2012 για τους δημοσιονομικούς κανόνες ε, που εφαρμόζονται στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης και απάλληψη κατάργηση του κανονισμού Ευρωπαϊκή Κοινότητα Euratom 1605 κάθετος 2002 που θα εφαρμοστεί από την 1η Πρώτου 13. Οπότε, Περί τίνος πρόκειται. Αυτές οι κατεξολόγηση, πράξεις πρέπει να ανακοινωθούν σε εσά τη συνεδρίασή μας σήμερα διότι λαμβανομένης υπόψη της συνθήκης το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις για αυτές τις εξουσιοδότηση πράξεις. Η προθεσμία γι' αυτό είναι δίμηνη. Και ήδη τρέχει. Ή θα αρχίσει να τρέχει. Άρχισε λοιπόν να τρέχει από τις 29 Οκτωβρίου όταν υπήρχαν όλες οι μεταφράσεις. Τότε και η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου που είναι αρμόδιες από τότε πρέπει λοιπόν με βάση τον, κανένα ε, με τον κανόνα 51 του ιστορικού μας κανονισμού μπορούν να ασχοληθούν με αυτές τις κατεξουδότης συμπράξεις. 29 Οκτωβρίου λοιπόν άρχισε να τρέχει αυτή η προθεσμία. Θέλει κανείς το λόγο. Α, η συγγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Η Σνάλφος Γκρέσλε. Παρακαλώ. Ο συντονίστρια εκπροσωπώ και τον Σνάλφο Ριβελίνη γιατί μου είπατε ότι είναι σε κάποιο αεροπλάνο με άγνωστο προορισμό. Ελπίζω ο προορισμός να είναι Βρυξέλλες. Να αναφέρω ότι το θέμα αυτό το συμφωνήσαμε με την Κομισιόν διότι οι κατεξουσιοδότητες πράξεις έχουν ήδη παίξει επανειλημμένα ρόλο. Να αναφέρω ένα θέμα θα ήθελα να κάνω μια συνεδρίαση με την ομάδα εργασίας γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι το θέμα της διαφάνειας. Δηλαδή να δημοσιεύονται οι ε, δικαιούχοι, αυτοί που λαμβάνουν καλύτερα επιδοτήσεις. Με βάση το άρθρο 21 που προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν ε, επιδοτήσεις από την Ένωση πρέπει να αναφέρονται στο, σε ένα site. Όμως μέχρι στιγμής η Κομισιόν δημοσιεύει μόνο τη χώρα που λαμβάνει τι επιδοτήσεις και όχι οι διευθύνσει συγκεκριμένε. Αυτό είναι υποχώρηση με βάση αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει. Πρέπει πραγματικά να υπάρξει πρόοδος. Τώρα λέγεται ότι όταν, εάν πρόκειται για φυσικά άτομα, τότε δημοσιεύεται η περιφέρεια σε επίπεδο οργάνωση του κράτους στο οποίο ανήκουν. Και σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία δημοσίευση. Σε μία περίπτωση που ξέρω για παράδειγμα, αναφερόταν όνομα και το κρατήδιο. Βάδι Βιρτεμβέργη. Χαντ Χέμπερ, Βάδι Βιρτεμβέργη. Αυτό είναι υποχώρηση. Διότι τσιχάνουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της διαφάνειας. Οπότε, να σας πω σαφώς, διότι αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα επίμαχο, είναι το μόνο που δημιουργεί προβλήματα από τις ε, εξουσιοδότηση πράξεις. Γι' αυτό θέλω βάσει το άρθρο 21 να το συζητήσουμε και με βάση το άρθρο 35 του Διεσημιακού Κανονισμού να το συζητήσουμε αυτό και αν θέλετε και αν συμφωνείτε να το συζητήσετε και θα ήθελα να προσκαλέσω μια συνεδρίαση τη ομάδα τι επόμενε δύο εβδομάδε. Θέλει κανεί το λόγο γι' αυτό. Λέω πρόεδρο, όχι. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σημαντική. Θέλει κανεί το λόγο. Ξέχασα κάποιον. Α, η Επιτροπή. Να ακούσετε τη γνώμη τη Κομισιόν. Μια που είστε εδώ, πείτε μα. Παρακαλώ. Ρωτάω την Κομισιόν. Δεν κατάλαβα ότι ήθελε το, η κυρία Γκρέσλε να μιλήσει κομισιόν, αλλά αν θέλετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πληροφορήθηκα ότι ο λόγος για την κατάσταση αυτή που σωστά περιέγραψε η κυρία Γκρέσλε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν επιτρέπει πληροφόρηση που επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ο λήπτης. Γι' αυτό η Κομισιόν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το επίπεδο NATS 2 αντί του 3 ή 4 για να είναι πιο δύσκολο. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Εάν γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα διατρέχαμε τον κίνδυνο το δικαστήριο να μας πει ότι δεν σεβόμαστε την απόφασή τους. Θα ήταν λοιπόν σωστό να το ξανασυζητήσουμε ειλικρινά το θέμα αυτό, ανοιχτά, για να ε, ε, αντιμετωπίσουμε τις ε, ε, βάσιμες ανησυχίες της κυρίας Γκρέσλε. Είστε ικανοποιημένοι κυρία Γκρέσλε. Όχι λέει η κυρία Γκρέσλε. Νομίζω ότι οι υποχωρήσεις, οι υπαναχωρήσεις είναι πάντα δύσκολη υπόθεση. Κοιτάξτε, Δεν θέλω να με κατηγορήσουν διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει που ασχολούνται με την διαφάνεια ότι δεν υποστηρίζω τι προσπάθειέ του. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια σύντομη συνάντηση να το συζητήσουμε αυτό. Εδώ μας λέει η Επιτροπή ότι απαγορεύεται να αναφέρονται συγκεκριμένα άτομα. Εγώ δεν βλέπω να αναφέρεται συγκεκριμένα, να, υπάρχει τέτοια απαγόρευση, να μας πει την άποψή του και ο υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρόεδρος. Βλέπουμε πόσο ε, επίμονη είναι η συγγήτριά μας, η συνεισηγήτριά μας, εντάξει, ευχαριστώ. Τελειώσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 3 στην ίδια αίθουσα. Τρεις ώρες ώρα. Διακόπτε τη